Colleagues, let's start with the next colleagues. We have one. Okay. Ah, yeah. <laughs> Thank you, Arno. Let's start with the next point of our agenda. Συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη, κατάστασης στο Σαχέλ. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον ειδικό μας ε, πρόσωπο για το Σαχέλ, τον επιστραμμένο για το Σαχέλ, τον κύριο Ματό, Παρακολουθούμε την κατάσταση στην περιοχή μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης στο Μάλι τον περασμένο Ιανουάριο του 2013. Οι συνάδελφοι που θα πάρουν το λόγο από την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ και σε θα μιλήσουν για το ρόλο της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θέλουμε να παρεμποδίσουμε την περαιτέρω κατάρρευση της χώρας στα πλαίσια της ισλαμιστικής και φονταμεταλλιστικής έντασης που επικρατεί. Η απόκριση όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν επαρκής, ειδικώ επειδή η πολιτική μας ασφάλειας και άμυνας στο Σαχέλ, όπως και εγκριθεί το, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2011, δεν υλοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Όμως, ευτυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέτεινε τη δέσμευση της για την ε, αποκλιμάκωση στο Μάλι και την όλη περιοχή. Οι πρόσφατες εκλογές στο Μάλι με τον πρόεδρο κύριο Κέτα, ο οποίος παρευρέθη στο Ευρωκοινοβούλιο το Δεκέμβριο, επέτρεψαν να έχουμε νέες δεσμεύσεις για την ε, διάθεση ανακοδόμησης και ανασυγκρότησης της χώρας. Ο πρόεδρος του Μάλι μας είπε ότι όλη η περιοχή πρέπει να προσπαθήσει για να διατηρήσει τη σταθερότητά τη μετά την, ε, τις αλλαγές στη Λιβύη αλλά και την υπόλοιπη, την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Συνάδελφοι, θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο τις αποστολές ε, της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας στην ε, περιοχή και να μας ενημερώσετε παρακαλούμε για την εκδίπλωση της στατικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαχέλ και συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά την ε, σύγκρουση, για την ε, δημιουργία ε, ισχυρών θεσμικών οργάνων στην περιοχή και για την ευρύτερη σταθεροποίηση της περιοχής. Κύριε Ντανζό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αντρέη. Καταρχήν τις ευχές μου. Καλή χρονιά σε όλους. Και θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη λύπη μας για τα δύο άτομα, ένας Δανός και ένας Βρετανός που επλήγησαν την προηγούμενη εβδομάδα από την απόπειρα, σκοτώθηκαν στην ε, απόπειρα, στην έκρηξη που έγινε σε ένα εστιατόριο στην Καμπούλ εμείς ε, πολύ συχνά επισκεφτόμαστε τις ε, ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται σε αποστολές και πολλές φορές συζητούμε για την ε, αποστολή τους χωρίς βεβαίως ποτέ να αμφισβητήσουμε τον επαγγελματικό χαρακτήρα και την αφοσίωσή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτίθενται όπως οι δύο ε, Ευρωπαίοι που σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Καμπούλ. Οι σκέψεις μας λοιπόν είναι με τις οικογένειές τους και βεβαίως η δέσμευσή τους, η αφοσίωσή τους είναι κάτι που μας υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα με τέτοιες αποστολές οι οποίοι πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους σε τέτοιες ε, μακρινές περιοχές. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Δεμοντό, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν ειδικό ε, απεσταλμένος και πρέσβης στο Μαλί. Φτάσατε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, εμείς βεβαίως είχαμε παρακολουθήσει και μας είχε απασχολήσει η κατάσταση στο Μάλι πριν ξεκινήσει αυτή η τελευταία κρίση και σκοπός μας είναι βεβαίως να υλοποιήσουμε τη στρατηγική των τριών τελευταίων ετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή, μια στρατηγική ανάπτυξης και ασφάλειας, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι έχει αποφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Μπορούμε μαζί σας να δούμε ποιος είναι ο απολογισμός αυτής της ε, πολιτικής, να δούμε ποιος είναι ο δικός μας ρόλος και στα πλαίσια των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις χώρες του Σαχέλ, αλλά και διότι μας εξέπληξε πάρα πολύ ο μεγάλος αριθμός των ειδικών απεσταλμένων ε, διαφόρων οργανισμών της ε, Αφρικανικής ε, Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Πρόντι και άλλοι. Τελικά αναρωτιόμαστε υπάρχει συντονισμός μεταξύ όλων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με όλους αυτούς τους οργανισμούς που δρούν επιτόπου και πέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Σαχέλ, που βεβαίως σήμερα επισκιάζονται από την κατάσταση στην Κεντρική Αφρική. Θα πρέπει ίσως να δούμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα την κατάσταση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, πώς βλέπετε τα πράγματα, πολλοί αναφέρονται σε ανασύσταση των τρομοκρατικών ομάδων εκτός της επικράτειας του Μάλι. Επικρατεί κάποια ανησυχία αυτές οι σκέψεις ευσταθούν, είναι δικαιολογημένες κατά την άποψή σας. Θα δικαιολογούσαν και μια στρατιωτική ενδεχομένως ε, επέμβαση στην περιοχή. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε την δική σας ε, αξιολόγηση και εκτίμηση, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτή η περιοχή απαιτεί μια ολοκληρωμένη και πιο γενική προσέγγιση, η οποία βεβαίως θα πρέπει να υλοποιηθεί. Περιμένουμε πολλά από αυτή την πολιτική και η δική σας εκτίμηση και παρουσίαση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για μας. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, σύσταση, την εξήγηση. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε υψηλό αξιωματούχο ή επιτετραμένο εκπρόσωπο, είναι πάντοτε σημαντικό να μπορεί να συζητήσει με εσά του ευρωβουλευτέ και να κατανοήσουμε πώ και εσεί αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, αλλά να ανταποκριθούμε και στι προσδοκίε σα σε διάφορου τομεί. Δείξατε πολλά ζητήματα ήδη με την πλούσια παρέμβασή σα. Καλύψατε πολλά θέματα. Εγώ είχα ετοιμάσει μια σύντομη ομιλία με σκοπό να θυμίσω κάποια στοιχεία. Νομίζω Βεβαίως το πιο σημαντικό θα ήταν να έχουμε διάλογο, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Ανακεφαλαιώνοντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε με μια πολύ καλή στρατηγική για το Σαχέλ. Ήμασταν από του πρώτου που είχαμε επινοήσει μια τέτοια συνεπή προσέγγιση ω προ την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή. Μα ακολούθησαν λίγο πολύ οι υπόλοιποι. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπή για, το, για την κατάσταση στο Σαχέλ μετά τι προσπάθειε σταθεροποίηση που ήταν θεαματικές το 2012. Φάνηκαν οι δυνατότητε τη διεθνού κοινότητα να κινητοποιηθεί και εντατικά με πολύ συγκεκριμένου κινδύνου ενώπιον τη. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε βρεθεί λίγο σε βαθιά νερά και έχουμε να κάνουμε με θέματα που είναι προβλήματα ουσίας, που είναι παρόντα στην περιοχή από δεκαετίες και που για το Σαχέλ είναι πολύ γνωστά. Λίγα λόγια λοιπόν για να ανακεφαλαιώσουμε. Το 2013 νομίζω ήταν μια χρονιά ορόσημο μετά την επίθεση των ομάδων του Βορρά που επιτέθηκαν στο υπόλοιπο τμήμα του Μάλι με την παρέμβαση της Γαλλίας, του ΟΗΕ και την ε, παραμονή της ε, CDAO με την ε, πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και με υψηλές φορολογίες. Έπειτα είχαμε μια πρώτη συμφωνία μετά μεταξύ της κυβέρνησης του Μαλή και των ένοπλων ομάδων του Βορρά στο Ουαγκαντουγκού και με την, υπό την αιγίδα της CDAO ώστε να οργανωθούν συνομιλίε ε, με τι ένοπλες ομάδε του Βορρά. Ήταν η πρώτη φορά που η διεθνή κοινότητα έπαιρνε θέση στο, στην ένοπλη σύραξη στη χώρα. Οι προεδρικές εκλογές ε, του προηγούμενου Ιουλίου-Αυγούστου διεξήθησαν σε κλίμα πολύ καλό, με μεγάλη νίκη, με ευρεία μάλλον πλειοψηφία, που επέτρεψε στον πρόεδρο να εκλεγεί ε, χωρίς αμφισβητήσεις. Πράγμα που δείχνει ότι η δημοκρατία στο Μαλί τελικά ήταν η πρώτη αντίδραση στην κρίση αυτή και η βασικότερη απάντηση. Οι βουλευτικές εκλογές ολοκληρώθηκαν τον ε, Δεκέμβριο, οπότε υπάρχει μια συνταγματική πλέον τάξη στη χώρα ε, και αυτό με την ευρεία συνένεση της διεθνούς κοινότητας, ιδίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μια μεγάλη σύνοδο που όλοι επιβεβαίωσαν την ε, συμφωνία του στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβριο στο Μαλί με τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανάπτυξη, την παρουσία του κ. Πίμπαλ τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης και εγώ μπόρεσα να συμμετάσχω. Επίσης υπήρξε σύνοδος του, του Συμβουλίου Ασφαλείας τον ε, Νοέμβριο με παρουσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά δεν είναι συνηθισμένα για την διεθνή κοινότητα. Να μπορέσει δηλαδή η διεθνή κοινότητα να εκδηλώσει τη βούλησή της και να μείνει συνεπής στη φτάση της. Αναντήρητα υπήρξαν κινήσεις πολύ αποφασιστικές και πέραν αυτό ε, υπήρξε ευρεία συνένεση, κάτι που επίσης δεν είναι ιδιαίτερα συχνό. Ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιώματα του ανθρώπου, η δημοκρατία ήταν ε, τα πρώτα, ε, οι πρώτες προτεραιότητες που μας απασχόλησαν για αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Έτσι δημιουργείται ένα νέο κλίμα, μια νέα κατάσταση. Εγώ τώρα επιστρέφω από ένα ταξίδι στη θάλασσα μεταξύ Μάλι, Αλγερίας και Μαυριτανίας και βλέπουμε ότι κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν ακολουθήσει μια αξιοθαύμαστη πορεία στην περιοχή, ιδίω ο που έχει μια πολιτική ανάπτυξης και ενοικοδόμηση πολύ εντυπωσιακή ε, με διάλογο με τη διεθνή κοινότητα ή η Μαυριτανία που πριν από λίγα χρόνια, χρόνια ήταν η πλέον ευάλωτη χώρα με πολύ συχνές επιθέσεις της Αλκάιντα στην επικράτειά τη, ενώ τώρα έχει καταφέρει να υλοποιήσει μια πολιτική ασφάλεια με συνειδητοποίηση του τι δράσει χρειάζονται ε, στα πλαίσια της μουσουλμανικής κοινότητας ώστε να μην υπάρχει πλέον ε, να μην υπάρχουν εντάσεις ή κίνδυνος εξτρεμιστικών εκδηλώσεων. Αυτέ οι εξελίξει είναι θετικές και δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν και θετικά αποτελέσματα. Τώρα από την άλλη πλευρά βρισκόμαστε σε μια περιοχή, γεωγραφική περιοχή που είναι μεταβατική, είναι ενδιάμεση. Έχει ευρύτερη διάσταση, έχει ευρύτερες διαστάσεις η κρίση αυτή, αφορά και περισσότερες χώρες, διότι ακριβώς οι αφρικανικοί φορείς είναι πολύ αδύναμη ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να τους ενισχύσουμε και πάντοτε ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν χώρο που βρίσκεται μεταξύ της Βόρειος Αφρικής και της, Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής. Το ζήτημα του Μαρόκου ε, περιπλέκει τα πράγματα διότι δεν συμμετέχουν στην Αφρικανική Ένωση. Υπάρχει λοιπόν πραγματικό πρόβλημα διαχείρισης στη σωστή κλίμακα, στην κλίμακα της πραγματικότητας αυτής της κρίσης. Κάτι που σημαίνει ότι δεν που δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτα. Η Αφρικανική Ένωση παίρνει και κάποιε πρωτοβουλίε που είναι όντω εύστοχε. Δημιουργήθηκε ένα Προεδρείο για το Σαχέλ, μια Επιτροπή για την Ασφάλεια. Η, η διαδικασία one shot στο πλαίσιο της άμυνας Βέβαια αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί ε, μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο στην ε, Μπάμακο ε, προβλέφθηκε να δημιουργηθεί ένας φορέας περιφερειακός για την συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, ώστε να καθορίσει κάποιες προτεραιότητες και κάποιους πρώτους στόχους τις ερχόμενες εβδομάδες, αλλά όλα αυτά ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί. Στο Μάλι Έχουμε να κάνουμε με ένα κράτο που ανέκαθεν ήταν ευάλωτο. Κάποιοι για να προκαλέσουν λένε ότι ουδέποτε υπήρξε πραγματικά οικοδομημένο και δομημένο κράτο στο Μαλή. Οι δυνατότητε των ε, θεσμικών οργάνων, των πολιτικών θεσμών ήταν πάντοτε περιορισμένε. Σήμερα υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε πολιτικέ που θα πρέπει να αναπτυχθούν, ιδίω για να υπάρξει μια σχετική αποκέντρωση στη χώρα αλλά ακόμη δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς, δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Υπάρχουν ενδιασμοί μεταξύ όσων μεταρρυθμιστών θέλουν μεγάλες αλλαγές, διότι λένε ότι θα πρέπει οι πολίτες να ξεχάσουν τα χρόνια της κρίσης και να ξεκινήσουν τις ε, εκβάθρων μεταρρυθμίσεις, αλλά τα πράγματα ακόμη είναι κάπως, ε, όλα γίνονται κάπως επιφυλακτικά. Πάντως σήμερα η κατάσταση στο βόρειο Μαλή είναι μια κατάσταση κάπως ε, αμετάλλακτη, δηλαδή πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις. Δεν υπήρξε πραγματικός αφοπλισμός, δεν υπήρχαν ε, πραγματικές εξελίξεις, συμβαίνουν ακόμη διάφορα δυσάρεστα. Ε, οι ξένες δυνάμεις, ή μάλλον οι τοπικές δυνάμεις, ο στρατός της χώρας ε, προσπαθεί να ενισχύσει το δυναμικό του αλλά με πολλές δυσκολίες. Η αποστολή του ΟΗΕ κάνει ό,τι μπορεί αλλά η εντολή που έχει από τη διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες επιτόπου. Τα πράγματα λοιπόν είναι αρκετά δύσκολα και ίσως και λίγο επικίνδυνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και παραμένει μια σχετική καχυποψία. Οι πρόσφυγε δεν θέλουν να επιστρέψουν στι αιστείε του, παραμένουν στη Μαυριτανία ή στην Μπουρκίνα Θάσο, διότι δεν υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών εθνικών κοινοτήτων. Ε, πρόκειται για μια επώδυνο ε, πραγματικά εμπειρία. Πολλοί είναι οι πρόσφυγε που μα έλεγαν ε, ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα. Αν κάποτε θα γυρίσουμε θα το δούμε, αλλά πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν η εθνική στρατηγική δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει καχυποψία μεταξύ των διαφόρων χωρών κιόλα. Η Αλγερία ε, είναι πάντοτε ένας καθοριστικός ε, παράγοντας στο όλο παιχνίδι, ο οποίος, ε, καθώς ο πρόεδρος της Αλγερίας πάντοτε έλεγε ότι ο βορράς του Μάλι, του Μάλι είναι ο νότος της Αλγερίας στην ουσία. Μιλάμε για μια χώρα πολύ δραστήρια στο διεθνές προσκήνιο, στην όλη περιοχή. Είδατε ότι τι τελευταίες μέρες η Αλγερία προσκάλεσε πολλέ ομάδες, ομάδες που στο Αλγέρι θα συζητούσαν για να βρουν μια λύση. Βέβαια δεν ήταν, κάποια, δεν ήταν κανένα φοβερό συμβούλιο, η διάσκεψη αυτή που οργανώθηκε στο Αλγέρι, αλλά υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ Μαρόκο και Αλγερίας για το Μάλι, για το Βόρειο Μάλι, για το Σαχέλ. Αυτό δεν είναι σίγουρα ένας πολύ καλός ιονός, γιατί μπορεί να προκαλέσει περιπλοκές ή εντάσεις. Οι τρομοκρατικές ομάδες σιγά σιγά να διοργανώνονται. Η γαλλική παρέμβαση βεβαίως γαλλικη παρεμβαση βεβαίω κέρια και κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού τους. Υπόθηκε περίπου το ίμιση των δυνατοτήτων των δημοκρατικών ομάδων. Οι ομάδες όμως μπορούν να αναδιοργανωθούν. Τις ερχόμενες εβδομάδες λοιπόν δεν θα είναι εντυπωσιακό αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα προστάσιο στη Λιβύη με δυνατότητες εκπαίδευσης, ε, εξοπλισμού. Θα μπορούσε να τραφοδητηθεί η ένταση στην περιοχή και οι τρομοκρατικές ομάδες στο βορρά του Μάλι σήμερα έχουν οργανωθεί πλέον σε δύο πόλους, την ΑΚΜΕ που είναι γνωστή και τον δεύτερο πόλο που είναι ακόμη πιο περίπλοκος, είναι πιο ε, διασκορπισμένος μεταξύ των διαφόρων ε, ομάδων του πληθυσμού και είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή και θα απειλήσει τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία διαθέτουμε, αλλά ο νότος της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μια, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτή τη κρίση είναι ακριβώ ο περίπλοκο χαρακτήρα τη. Ξεκινήσαμε από μια κρίση στο Σαχέλ και τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σαχέλ, εντοπίζοντα το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Ήγηρα ω τι τρει χώρε προτεραιότητα. Και βλέπουμε ότι τελικά καλύπτεται όλη η περιοχή ε, του Σαχέλ. Δεν θα φτάσουμε στο Σουδάν γιατί εκεί υπάρχουν ειδικέ προτεραιότητε, αλλά και οι χώρε του Μαγκρέμπ ε, επηρεάζονται από το Σαχέλ ή ο νότος της Λιβύης. Μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που αφορά το Σαχέλ και τη Σαχάρα, χωρίς να περάσουμε μέχρι τη Σαχάρα βέβαια και να τη διασχίσουμε, αλλά από πολιτικής άποψης είναι χώρα που αφορά τα κράτη του Σαχέλ, ε, της, ε, του Μαγκρέπ, της Βορείου δηλαδή Αφρικής και πολλά κράτη της Δυτικής Αφρικής. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανεί μια τέτοια κρίση. Ε, περιλαμβάνει αναπτυξιακές παραμέτρους, ε, μεσοπρόθεσμε, μακροπρόθεσμε, με μια δημογραφική εξέλιξη εκρηκτική, με ε, διαστάσεις ασφάλειας, οικοδόμηση κρατών και το πώς είναι αλληλένδετοι και πολύπλοκοι, περιπλέκονται μεταξύ τους αυτοί οι παράγοντες. Μια κρίση λοιπόν που είναι δύσκολο κανεί να την περιγράψει, να την αντιληφθεί και να την αναχαιτήσει. Πάντως, Έχω εργαστεί επί επιμακρών ε, ε, σε αυτά τα κράτη και ε, νομίζω ότι γνωρίζω καλά ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες, γι' αυτό και τόσες οι δυσκολίες της διεθνούς κοινότητα να αντιμετωπίσει την κρίση. Εδώ το θέμα είναι πόσο θα καταφέρουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά, διότι αποφασίζουμε να αφιερώσουμε κάποια κονδύλια, θέλουμε οι αλλαγέ να γίνουν γρήγορα και να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα, όμω στι χώρε του Σαχέλ δεν συμβαίνουν τα πράγματα τόσο αυτόματα όσο θα τα θέλαμε. Για μια κρίση ιδίω τόσο περίπλοκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε παρούσα στο, στη διάρκεια όλη αυτή τη περίοδου Τη κρίση, ξέρετε τι διάφορε διαστάσει τη παρέμβασή μα. Νομίζω ότι ιδίω φέτο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια εδραιώσαμε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνέ προσκήνιο. Το ψήφισμα του ΟΗΕ για το οποίο ήμουν υπεύθυνο ω ειδικό επιτεταμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ψήφισμα αυτό στον ΟΗΕ, είναι κάτι που παροτρύνει όλου να συνεργαστούν και σε διεθνές επίπεδο η CDO, ε, η Αφρικανική Ένωση, η ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμαστε στενά για τα θέματα αυτά σε όλα τα δυνατά επίπεδα και νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά έχει καταλάβει τη θέση που της αρμόζει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει πολλέ πρωτοβουλίε πρόσφατα. Η πιο θεαματική ήταν η διάσκεψη των Βρυξελών για το Μάλι, με, με προτεραιότητα να σταθεροποιηθεί το κράτο, να κινητοποιηθεί η διεθνή κοινότητα για τη σταθεροποίησή του. Ήταν ε, πολύ σημαντική και η στήριξη από του ίδιου του υπευθύνου του Μάλι. Στο βορρά επίση τη χώρα προβλέψαμε χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από μη κυβερνητικέ οργανώσει είτε από φορεί του ΟΗΕ. Υπάρχει σημαντική δημοσιονομική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μάλι για σωστή ρύθμιση των δημοσιονομικών τους με την παρουσία του Διεθνούς Ταμείου και εκεί υπήρξαμε παρόντες. Υπήρξαν επίσης κάποιες αποστολές της ενιαίας πολιτικής ε, ασφαλείας και η PCM η οποία ε, κατάφερε να δώσει αποτελέσματα. Η EUCAP η οποία είχε σημαντικές πολιτικές επιτυχίες και κατάφερε και αυτή να καθορίσει συγκεκριμένες πρακτικές για την επιχειρήσή της και η UBAM, η οποία προβλέπει συγκεκριμένες επιχειρήσεις και μάλιστα επιτυχημένες. Τώρα για, τον, ε, ε, για, την, προ, πρόνοια κατά της ρίζος, ρίζος παστικοποίησης, αυτή ήταν μια πιο περίπλοκη προσπάθεια, αλλά λόγω της πρωτοτυπίας της του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, πετύχαμε και εδώ κάποια πράγματα. Ε, για τον προγραμματισμό του επόμενου Fed. προβλέψαμε τον συντονισμό των διαφορών υπηρεσιών και υπεύθυνων ομάδων εργασίας. Η περιοχή του Σαχέλ χρησιμοποιήθηκε ως πλαίσιο καθορισμού πολιτικών για τα ερχόμενα χρόνια με πολύ συγκεκριμένες αναφορές, με πολύ ακριβείς λεπτομέρειες και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία επικαιροποίηση της στρατηγικής για το Ροσαχέλ η οποία έχει δημιουργηθεί πριν από τρία χρόνια. Λογικό ήταν κάποια στιγμή να ενημερωθεί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις συζητήσεις μας με τις διάφορες ομάδες που είναι υπεύθυνε για το Μάλι την Μαυριτανία. Από την κρίση λοιπόν αυτή αντλήσαμε το εξή συμπέρασμα, ότι από κοινού πρέπει να καθορίσουμε που θέλουμε πραγματικά να οδεύσουμε και σε αυτή τη στρατηγική. Δεν μπορώ να περάσω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά για να δώσω μια απάντηση και σε αυτά που είπατε εσείς Πρόεδρε για την διεθνή συνεργασία πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα περίπλοκο. Στο Μάλι, στο Σαχέλ έχουμε μια από τις καταστάσεις όπου μια από τις περιπτώσεις που τα πράγματα δεν έχουν πάει και τόσο άσχημα. Έχουμε και κάποια προηγούμενα βεβαίω. Υπήρχε ήδη ένα σύστημα διεθνούς συνεργασίας που είχε δημιουργηθεί στην ε, Αμπάμακο σιγά σιγά. Εγώ ίδιος είχα εργαστεί για τα θέματα αυτά τα προηγούμενα χρόνια τα πράγματα έχουν πάει σχετικά καλά λοιπόν. Παρ' όλα αυτά πολλές χώρες, πολλοί φορείς δεν θέλουν να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού. Άρα όταν μιλάμε για τον συντονισμό όλοι είναι ενθουσιώδεις όταν μιλάμε για τον συντονισμό των άλλων αλλά όχι για τον εαυτό τους. Δεν θα δώσω παραδείγματα προσωπικά, αλλά πραγματικά δεν έχουμε και φοβερό περιθώριο ελιγμών εδώ. Η συνολική μας προσέγγιση πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μακρόν. Η στρατηγική μας για το Σαχέλ ε, δείχνει πραγματικά ότι έχουμε βούληση για μια ε, συνολική προσέγγιση. Η διάρθρωση των προσπαθειών μας στην ασφάλεια και την ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει βεβαίως ανάλογα με την βούληση που υπάρχει και επιτα, σίγουρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες που εμπλέκονται. Κάποιε φορέ κινητοποιούνται προβολικά πολλοί φορεί στα πλαίσια του ίδιου οργανισμού, ε, πολλά διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίε, το ίδιο και στις χώρες. Μη κυβερνητικές ε, φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, Όσο περισσότερο συντονισμό απαιτείται, τόσο πιο δύσκολο είναι να υπάρξει συνοχή στι ε, προσπάθειε Εδώ ε, νομίζω ότι έχουμε παρόλα αυτά περάσει από πολύ ενδιαφέροντα στάδια στην όλη διαδικασία και υπάρχει μια κοινή θεώρηση, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, μια κοινή θεώρηση η οποία σιγά σιγά αποκρισταλώνεται. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσει, ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα, είναι η συνεργασία μας με τα κράτη αποδέκτες, ε, ε, όπως το Μάλι η σχέση μεταξύ των χωρών αποδεκτών δικαιούχων, δηλαδή όσων είναι δικαιούχοι της διεθνούς βοήθειας και των ε, δωρητών, είναι πολύ πιθανό οι δικαιούχοι να δέχονται με μεγάλη χαρά την βοήθεια, αλλά όχι το ίδιο και τα επικριτικά σχόλια. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια της εταιρικής μας σχέσης να καθορίσουμε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, την καλύτερη δυνατή πρωτοβουλία ή πρακτική που να εφαρμόζεται. Η περίπτωση του Μάλι, όπω είπα προηγουμένω, είναι περίπλοκη, διότι πρόκειται για μια από τι χώρε που βοηθήθηκε από τη διεθνή κοινότητα επί μια εικοσαετία περισσότερα από πολλέ άλλε, αλλά είναι και μια χώρα που είχε πολύ συγκεκριμένε δυσκολίε. Κάτι που δεν πήγε καλά. Τι ήταν αυτό, ήταν ότι ίσω δεν καταλάβαμε και δεν αντλήσαμε τα σωστά διδάγματα από τον διάλογο που δεν είχαμε με το Μάλι. Οπότε θα πρέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να θέσουμε σωστότερα ερωτήματα για τις συνθήκες επιτυχίας της διεθνούς δράσης σε τέτοιου είδους χώρες. Υπάρχει λοιπόν ε, η ανάγκη να εντοπίσουμε μια σωστή ισορροπία γιατί κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Το αν θα έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο τώρα, δεν το ξέρω. Η διάσκεψη των Βρυξελών ήταν ε, μια υπόσχεση βοήθεια για το Μαλί πολύ σημαντική, 3 δις ευρώ, αλλά 3 εκατομμύρια ευρώ μάλλον, αλλά τώρα το αν η των 3 εκατομμυρίων ευρώ θα συνοδευτεί από σταθεροποίηση στην περιοχή δεν το ξέρω. Θα πρέπει να έχουμε καθημερινή επαφή με τους διάφορους συνομιλητές μας. Κάποιες φορές δεν έχουμε τη διάθεση να λέμε και να επαναλαμβάνουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Μιλάμε για μια διαδικασία και διπλωματικού χαρακτήρα, με δισταγμούς, με όλα τα σχετικά ρίσκα. Ίσως και δύο λόγια για το δικό μου τον ρόλο. Εγώ ξεκίνησα το Μάρτιο. Στην ε, ομάδα μου έχω τέσσερις συνεργάτες Ξεκινήσαμε όλοι μαζί από το Σεπτέμβριο, είμαστε δηλαδή καινούργια σχετικά ομάδα και ήμουν ε, παρόν στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Ο δικός μου ρόλος λοιπόν ε, λειτουργεί ικανοποιητικά. Ο τρόπος που με δέχτηκαν οι χώρες, οι κυβερνήσεις ήταν πολύ καλός. Ε, γιατί ήταν πολύ θετικό το ότι οι ευρωπαϊκές αρχές, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφάσισαν να παρέμβουν περισσότερο, πιο ενεργά στην περιοχή αυτή. Εργάστηκα λοιπόν ιδιαίτερα για την επίλυση αυτής της κρίσης στο Σαχέλ. Πρέπει να σας πω ότι επισκέπτομαι αυτές τις χώρες, αυτούς τουλάχιστον που με καλούν, προσπαθώ να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, παρακολουθώ αυτά που συμβαίνουν, αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανταλλάσσω απόψεις με όλους τους ε, παρεμβαίνοντας καθώς και με την ε, ύπατη βεβαίως ε, πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής καθότι όλοι εργαζόμαστε υπό τη δική της αιγύρα. Σήμερα πρέπει να πω ότι τα πράγματα περιπλέκονται είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η συνοχή της Διεθνούς Κοινότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και πρέπει να δεχτούμε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει και ότι η αποτελεσματικότητα ίσως δεν φαίνεται ακόμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Βεβαίως πολλά περιγράψατε, αλλά είναι και περίπλοκος ο ρόλος σας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ασφάλεια και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Αναφερθήκατε στο επιχειρησιακό κομμάτι των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Νίγηρα και στο Μάλι. Επισκεφτήκαμε αυτή τη χώρα πέρσι εμείς. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσουν και σε κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει ανάγκη, υπάρχουν ε, από μέρους άλλων χωρών ε, αιτήματα για να εξάγουμε το ίδιο μοντέλο επιχείρησης, επέμβασης και κάπου αλλού. Ο κύριος Γκάλερ όμως έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πολύ σωστά είπατε. Με ακούτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε στην περιπλοκότητα της όλης περιοχής και ήδη το 2011 θεσπίστηκε η στρατηγική για την περιοχή του Σαχέλ. Βασιστήκαμε σε μια ανάλυση, ξέραμε πόσο ευαίσθητη είναι η όλη περιοχή και προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε ανάλογα με αυτά που ξέραμε. Δεν θέλω τώρα βεβαίως να κάνω ανασκόπηση του παρελθόντος. Η ερώτησή μου αφορά πιο πολύ στις ένοπλες δυνάμεις που ενδεχομένως θα στείλουν τα αφρικανικά κράτη, η Αφρικανική Ένωση. Τι στοιχεία έχετε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αλλά και τη χρηματοδότηση τέτοιων αποστολών. Το African Peace Facility έχει προβλεφθεί να σταλούν κάποιες ε, ενοπλές δυνάμεις αφρικανικών χωρών υπάρχει καλή συνεργασία με τις δικές μας αποστολές. Υπάρχει συντονισμός, ε, ποιος κάνει τι. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει καμία προϊστορία συνεργασίας, καμία εμπειρία. Και κατά κάποιο τρόπο κινδυνεύουμε εδώ να βρεθούμε σε μια τελείως αναποτελεσματική ε, αποστολή στο Μάλι η νέα κυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στην ε, σταθερότητα και όσον αφορά το κράτος δικαίου αλλά και όσον αφορά την κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας, της αστυνομίας και όλες της διοίκησης. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τι κάνουμε επί τόπου. Τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους ανεξάρτητα και τι πρέπει να τους βοηθήσουμε να κάνουμε. Η αναγκόμες. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη για την περιγραφή της κατάστασης. Σημείωσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα όμως που θέλω να σας θέσω είναι τι παραπάνω μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά που κάνει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος ε, στους υπουργούς μας, διότι έχουμε να κάνουμε με μία μείζωνα κρίση. Και σε γειτονική περιοχή. Μείζωνα κρίση, λοιπόν, που δεν αφορά μόνο τους θεσμούς και τις χώρες της περιοχής εκείνης, αλλά και την ασφάλεια των δικών μας πολιτών. Γιατί οι τρομοκρατικές οργανώσεις που εδράζονται εκεί δεν έχουν μόνο τοπικούς στόχους, τοπική δράση. Μπορεί να θέλουν να ξαπλώσουν τη δράση τους. Τι περιμένουμε εμείς τώρα. Περιμένουμε να υπάρξει μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση για να συγκεντρωθεί το μυαλό των ε, υπουργών μας και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Τι περιμένουν, δεν καταλαβαίνω. Ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα έγινε με καθυστέρηση, ακόμη και σε σχέση με τη στρατηγική που είχαμε θεσπίσει εδώ και καιρό. Είχαμε μάλιστα το πίσω και απειλές. Πάρα πολύ λίγα πράγματα έγιναν και με πάρα πολύ λίγο συντονισμό. Είπατε ότι υπάρχει δυσκολία για όσους δεν θέλουν να συντονιστούν σε επίπεδο διεθνών οργανισμών. Εμείς συντονιζόμαστε. Έχω το παράδειγμα της Λιβύης να σας αναφέρω. Πολύ σωστά αναφέρατε τον πολύ ξεκάθαρο σύνδεσμο και σχέση που υπάρχει με όλο αυτό το χάος στη Λιβύη. Τελικά τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συντονιστούν μεταξύ τους και δεν κάνουν και τίποτα ε, προς αυτό το στόχο. τα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Επίσης, επειδή μιλήσατε για τη σημασία παραγόντων όπως η Αλγερία, το Μαρόκο. Κράτη σημαντικά που όμως όχι μόνο δεν έχουν ρυθμίσει τα βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη Σαχάρα και που βοηθάει και η Ένωση να τα σπρώξουν κατά το χαλί, αλλά πώς να το πω τώρα, προχωράνε, επεκτείνονται και στο Μάλι τώρα. Βόρεια, στο βόρειο μου. Είχαμε εκπροσώπους, μια αντιπροσωπεία ε, που δεν ξέρω, φαίνεται να υπάρχει μια άρνηση από πλευράς Μάλι ότι στο Βόρειο Μάλι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι πρέπει να, γίνει, να, να βρεθεί κάποια διευθέτηση με τον πληθυσμό. Και όλα αυτά βέβαια είναι βούτυρο στο ψωμί των τρομοκρατών. Είπατε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα Αλγερίας Μαρόκου και αυτή τη βλέπουμε να φτάνει μέχρι το βόρειο Μάλι. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικά. Μπορούμε να συνεχίσουμε να βάζουμε κάτω από το χαλί όπως και με τη Δυτική Σαχάρα αυτό το πρόβλημα. Merci. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για αυτό το πρόβλημα διεθνού συντονισμού. Φαντάζομαι το ζήτημα είναι και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο σημαντικότερος ε, παράγοντας, πρωταγωνιστής που Έχουμε την Αφρικανική Ένωση, έχουμε τον ΟΗΕ ή μήπως υπάρχει προσδοκία αυτό το κράτος που έχει καταρρεύσει να γίνει ένα είδος προτεκτοράτου κάποια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μου πείτε και την δική σας προσωπική άποψη σε σχέση με την ε, συνεκτικότητα της απειλής ε, σε όλο το Σαχέλ. Διότι αντιλαμβανόμαστε αυτό το αυτά τα franchises που αναπτύσσονται, τις συνεργασίες, τις σχέσεις αυτές. Εσείς μιλάτε με μέλη των επαναστατημένων, εξεγερμένων ή των ανταρτών. Τι θέλουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους, είναι κάτι επιφανειακό ή κάτι άλλο τρέχει. και υπάρχει αυτή η δαιμονοποίηση, η δημιουργία ενός μύθου που εμείς ουσιαστικά φτιάξαμε. Ποια είναι η πραγματικότητα. έρχονται και φεύγουν ε, αυτές τις ενότητες εκεί επί τόπου που έχουν συγκεντρώσει τις πάνε και τις πάνε μετά κάπου αλλού. Κύριος, η κυρία Λέζιν και μετά ο κύριος Τάνοκ. Ja, vielen Dank äh, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Καλύψατε πάρα πολλούς τομείς. Θα ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά δεν νιώθω πιο έξυπνη από όσο ήμουν πριν έρθετε. Τι να σας πω, είπατε πράγματα αρκετά ασαφή και θυμάμαι ότι η λέξη περίπλοκο, η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού, αυτές είναι έννοιες που έχουμε ακούσει και ξανακούσει. Επίσης μιλήσατε για πολλά σχέδια τα οποία είναι πολύ καλά και θα ήθελα να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν μιλάτε για σχέδια και προγράμματα, τι είναι προγράμματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, στρατιωτικά, απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό, πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αξιολογήσουμε για τι προγράμματα πρόκειται και ποιος είναι ο σκοπός τους. Στη Γερμανία διαβάζω στον τύπο ότι θα υπάρξει ενδεχομένως και γερμανική συμμετοχή στην αποστολή του Μάλι. Διαβάσαμε πολλά πράγματα επίσης για την κοινή αποστολή της Γαλλίας και της Γερμανίας και ότι επιτέλους, επιτέλους θα υπάρξει και μία πραγματικά ευρωπαϊκή αποστολή. Τελικά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για δύο χώρες που από κοινού θα στείλουν δυνάμεις στο Μάλι. Πρόκειται για αποστολή ευρωπαϊκή που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε αυτή την αποστολή και τελικά ποιος είναι και ο πραγματικός σκοπός αυτής της επέμβασης στο Μάλι. Η κυρία Γκόμες είπε πολύ συγκεκριμένα ότι ναι, στην περιοχή υπάρχουν τρομοκράτες. Πολύ συγκεκριμένα όμως από στρατιωτικής απόψεως θα ήθελα να μου εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται. Γιατί όταν μιλάμε για τον πόλεμο του Αφγανιστάν σκεφτόμαστε αμέσως τρομοκράτες. Τα αποτελέσματα μπορείτε να μου πείτε στην πράξη ποια είναι ή ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το Μάλι. Τι μπορείτε, αν θέλετε, να μας ε, πείτε επιτόπου για την επέμβαση και τα αποτελέσματά της στο Μάλι. Τσάλ Στάνοξ, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, συγχαρητήρια. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που αναλαμβάνεται σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Ο Στίβεν Ομπράιαν ήταν ε, ο ειδικός απεσταλμένος από το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή και αυτό δείχνει βεβαίως ότι και άλλες χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την περιοχή και όχι μόνο η Γαλλία. Πρόκειται για μια κρίση η οποία βεβαίως πλήττει όχι μόνο αυτή την περιοχή της Αφρικής αλλά και τον Νότιο Σουδάν και την Κεντρική Αφρική. Και θα ήθελα να εξετάσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα μέρη της Αφρικής. Νιώθετε ότι σήμερα έχει μειωθεί λίγο ο ενθουσιασμός των Ευρωπαίων όσον αφορά την στήριξη αυτών των αποστολών, αυτών των επεμβάσεων και όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα αλλά και όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Για πείτε μου, τρομοκράτες είναι αλήθεια ότι βελτιώνουν την συνεργασία τους και τον συντονισμό τους και στη Σομαλία και στην Αλγερία αλλά και στην περιοχή του Σαχέλ, Μάλι λοιπά Αποτελούν μια πραγματική απειλή για την ασφάλειά μας. Επίσης όσον αφορά τις ομάδες τρομοκρατών της Συρίας, Τζιχάτ και άλλες στην Σαουδική Αραβία, ποιο είναι ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και ενδεχομένως ε, της Τουρκίας όσον αφορά τις ομάδες αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Συρία. Ναι, και όχι μόνο στη Συρία, απειλούν και έξω, μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. διότι η χρηματοδότηση, τα όπλα και οι αγωνιστές, οι τρομοκράτες φεύγουν από αυτή την περιοχή και από τη Συρία και φτάνουν μέχρι την Αφρική. Τι έχετε να πείτε εσείς και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης, τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι έχουν καλύψει ουσιαστικά τα βασικά με ερωτήματα. Όμως, και στην παρέμβαση του πρέσβη και στη συζήτηση, βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει απειλή, κίνδυνος, πραγματικός κίνδυνος τρομοκρατίας από την Αλκάιντα και τις διάφορες παραλλαγές της και παρακλάδια της. Δεύτερον, βλέπουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, δεν το κάνει βέβαια τώρα, κατά πόσον αρκεί έχει οριστεί επαρκώς μάλλον η δράση της ε, στην περιοχή είναι ένα άλλο θέμα, πρέπει όμως να το κάνει και γιατί το λέω αυτό. Για τις άλλες περιπτώσεις στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα ε, κατά πόσο θα πρέπει να είναι ένας διεθνής πρωταγωνιστής Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της ασφάλειας εμείς θεωρούμε ότι έχει ένα ρόλο. Γιατί. Πρώτον γιατί απειλείται άμεσα και από πολιτικής και από γεωγραφικής πλευράς και από δημογραφικής πλευράς από τρομοκρατικά στοιχεία της περιοχής αυτής. Τρίτον, αυτό που λέγατε. Αρκεί ή δεν αρκεί. Από τα λόγια που είπα, το πως είπε και μια συνάδελφος, δεν συνάγουμε ακριβώς ε, πού έγινε οι αδυναμίες, ε, οι ελλείψεις και τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για να είναι πιο ορατή δράση και πιο προβεβλημένη. Διότι πραγματικά δεν θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις και μετά να δράσουμε πιο αποτελεσματικά. Και όλο αυτό βέβαια εντάσσεται σε ένα στρατηγικό όλο, σε ένα στρατηγικό πλαίσιο που περιλαμβάνει, πολύ σωστά το είπατε, την ασφάλεια τη περιοχή, την ανάπτυξη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά, Όμω εγώ θα ήθελα να σα υποβάλω δύο ερωτήματα. Τα υπόλοιπα τα έθεσαν οι προλέσαντε συνάδελφοί μου. Πρώτο ερώτημα. Δεν είναι τόσο επιχείρηση όσο ένα πρόγραμμα, μια αποστολή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κράτον μελών της ή δεν συμφωνούν με αυτήν την αποστολή κάποια κράτη-μέλη. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα κράτη-μέλη του Νότου. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, ενστερνίζεται αυτή τη την δράση, αυτή την αποστολή. Και δεύτερον, δεν άκουσα στη δική σας παρέμβαση, σε κάποια άλλη παρέμβαση, να γίνεται μνήα σε μια δύναμη που πάντοτε αναφέρει στα διεθνή ζητήματα ή τι είπα. Δεν αναφέρθηκε. Τι κάνουν οι ΗΠΑ, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν μια δική τους αποστολή. Μέχρι τώρα ήταν ένα στοιχείο κλειδί οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διεθνείς ε, δράσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν κατά πόσον αφήνουν τη διεθνή κοινότητα εκπροσωπούμενη από τα Ηνωμένα Έθνη και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ, Λέω ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρον βλέπετε κύριε Πρέσβη, δείχνει η Επιτροπή μας για το θέμα του Σαχέλ. Ξέρω ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμά μας, η ημερήσια διάταξη έχει πολλά σημεία, σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν καλύτερα στα πολλά ερωτήματα. Τρεις ε, βασικές σκέψεις ε, συγκράτησα που ομαδοποιούν ε, και κάποια από τα σημεία που αναφέρθηκαν. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μια από τις δυσκολίες της διεθνούς δράσης είναι οι σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών, κυρίαρχων οντοτήτων. Ως παράγοντες, ως πρέσβης, πολλές φορές είδαμε υπουργού, πρωθυπουργού, προέδρους και τους είπαμε, ξέρετε κάτι δεν πηγαίνει καλά, θα μπορούσατε να λάβετε την τάτη, την απόφαση, να είστε προσεντάτε τη δίνα κατεύθυνση. Δεν ε, συμβαίνει πάντοτε ένας πρέσβης ή ένας ε, σύμβουλος να εισακούεται. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν συνεχώς τέτοιου είδους ε, ζητήματα. Γνωρίζουμε ότι είναι κυρίαρχες οι χώρες αυτές και είναι και πραγματική πρόκληση για κάποιες από αυτές τις χώρες η απόκτηση και διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας. Προσπαθούμε να πετύχουμε αποτελέσματα, πολλές φορές όμως ε, δεν το καταφέρνουμε. Δεύτερον, αποτελεσματικότητα τη διεθνού βοήθεια, αναπτυξιακής βοήθεια, διεθνού δράσης. Και αυτό παραμένει μείζον ζήτημα. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει. Η ΟΣΑ κάνει τι συστάσεις της, αλλά πάρα πολλά προβλήματα παραμένουν. Προκλήσεις σημαντικέ. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι η κλειδί είναι μια πιο στενή εταιρική σχέση η βελτίωση και ενίσχυση ε, της οικοδόμησης κράτους και πολύ μεγάλο μέρο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε εκεί ακριβώς οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ένα πλαίσιο, δεν έχουμε ένα συνομιλητή και επομένως η αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας δεν είναι ε, στο ύψος των προσδοκιών μα. Ε, οι διάφοροι υπάλληλοι, οι ψηφιακές οργανώσει κτλ. προσπαθούν να δράσουν, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά είναι λίγο σχετική η όλη προσπάθεια. Και έπειτα έχουμε και την όλη περιοχή στο Σαχέλ. Περιφερειακά είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει και διασυνοριακή όμως ε, προσέγγιση που διέπεται από μια παραδοσιακή αντιμετώπιση από όλα αυτά τα κράτη που βασίζουν όλα στην κυριαρχία τους. Έτσι βλέπουν τα πράγματα. Υπάρχει μια μικρή ε, άτολμη πρόοδος, κάποιες χώρες συνεργάζονται, δύο χώρες μαζί μας συνεργαστούν, αλλά τέλος πάντων έχουμε πολλά προβλήματα ακόμα. UTM, UCAP ε, ναι, συνάγουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο κάπου αλλού. Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει κατά παραγγελία να είναι εξατομικευμένες οι επιχειρήσεις και οι αποστολές μας έκαναν τη διαδρομή τους αυτές οι δύο επιχειρήσεις. Οι αποστολές είχαν τα καλά, τα κακά τους σημεία βελτιώθηκαν. πάντων, δεν νομίζω ότι υπάρχουν στην ε, περιοχή χώρε που θα ζητούσαν σήμερα μια αντίστοιχη επιχείρηση. Εγώ γύρισα μόλι από την Μαυριτανία. Οι αρχέ τη χώρα ε, θα ήθελαν κάτι που να αποκρίνεται καλύτερα στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα κατά κάποιο τρόπο. Ορισμένες φορές αυτό δημιουργεί ζητήματα, είναι λίγο λεπτό το θέμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Οι χώρες αυτές πιο εύκολα συνεργάζονται με κράτη-μέλη όπως είναι η Ισπανία ή η Γαλλία που, που δραστηριοποιούνται περισσότερο. Και όχι συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε βρει ε, τον τρόπο εργασίας, ε, τον ιδανικό ακόμη επιχειρησιακό σκέλος, ε, στρατιωτικό. Αυτό που ξέρουν να κάνουν ε, οι στρατιωτικοί είναι αυτό που κάνουν. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολο, κάποιες φορές όχι. Και εξαρτάται από το στράτευμα. Με άλλους τα πάμε καλύτερα, με άλλους λιγότερο. Τώρα η χρηματοδότηση απευθείας ε, από την Ένωση δεν υπάρχει. Στη ΜΙΣΜΑΡ είχαμε μία έμεση χρηματοδότηση, δηλαδή χρηματοδότηση οργανώσεων, αλλά δεν ε, χρηματοδοτούνται οι δυνάμεις συμμάχοι στα στρατεύματα αν μπορώ να το πω έτσι. Και μετά υπάρχει και το θέμα του επαγγελματισμού. Επιτόπου καλά πηγαίνουν τα πράγματα πάντως. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό ρόλος των κοινοβουλίων των χωρών. Δεν είναι επαρκή, σαφές και θα πρέπει να ενισχυθεί διακυβέρνηση στο κράτος δικαίου για αυτόν τον λόγο. Έχουμε ανοιχτά συστήματα παντού σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία ή το διάλογο, αλλά συχνά υπάρχει με αντιπολίτευση η οποία δεν έχει πολύ δύναμη, η εκτελεστική εξουσία είναι στα χέρια του Προέδρου και το Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ πιο αδύναμο ρόλο σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε σήμερα να έχει δεν είναι επάρκε οι κριτικέ του ικανότητε. και δυνατότητε. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να έχουμε μια πιο συνεκτική δημόσια πολιτική. Τι μα δυσκολεύει σήμερα στι προσπαθίε μα για ενίσχυση της ασφάλειας. Το ότι οι χώρε δεν έχουν ακόμη μια απόλυτα συνεκτική και πλήρη πολιτική ασφάλεια. Μέσα ασφάλεια υπάρχουν, έχουμε εθνοφυλακή, στρατό, αστυνομία, αλλά δεν υπάρχει απόλυτα συντονισμό με συγκέντρωση και πραγματοποίηση των μέσων. Υπάρχουν ανεπάρκειες και τα προβλήματα τα βλέπουμε λίγο πολύ παντού. Δημόσιες εξουσίες πρέπει να ενισχυθούν, οι πολιτικές οι δημόσιες πρέπει να εφαρμόζονται και βέβαια με διάλογο και με συνεργασία με τα κοινοβούλια γιατί εκεί γίνεται πολλή δουλειά. Τώρα για τη Δυτική Σαχάρα. Ε, με ξεπερνάνε λίγο αυτά που αναφέρατε. Η διεθνής κοινότητα έδωσε ε, στη ΣΥΠ υπάρχει και ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα, ο κ. στον συνάντησα μάλιστα, ο οποίο χειρίζεται αυτό το θέμα. Εκεί έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα μάλλον μέχρι στιγμή. Τώρα, εγώ προσωπικά έχω την πεποίθηση ότι ο πολιτικό διάλογο. η διπλωματική και πολιτική δράση τη Ένωση, απέναντι σε όλε τι χώρες τη περιοχή μπορεί να ενισχυθεί. Αυτό είναι και ο ρόλο μου και ίσω. Ε, ως και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Πρέπει ε, να έχουμε μεγαλύτερη βαρύτητα ως πολιτικοί πρωταγωνιστές, πρέπει να εδραιώσουμε το ρόλο μας και στον τομέα της ασφάλειας. Αλλά αν έχουμε ανάπτυξη, ε, πολιτικό σκέλος και ασφάλεια, το τρίτο σκέλος, το πολιτικό είναι αυτό που πρέπει να ενισχύεται. Δεν είναι εύκολο αυτό γιατί η διπλωματία σιγά σιγά αναπτύσσεται. Κάποιες φορές είναι δύσκολο, κάποιε φορές λιγότερο δύσκολο, άλλοτε συνεννόμαστε καλύτερα με κάποιον εταίρο, άλλοτε όχι. Και ενίοτε δημιουργούνται προβλήματα, έχουμε κάποια συμβάντα. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει απαιτούμενη βούληση για την επίλυση των προβλημάτων και ότι δεν διακυβεύονται συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα για τις τρομοκρατικές ομάδες σήμερα ε, ποικίλουν ε, λίγο πολύ γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες, ε, την ΑΚΜΗ τη γνωρίζετε. Είναι σαν σέκτα. Στρατιωτικοποιημένη, επιθετική, φονταμεταλιστική, το Μουζάο πιο πολύ κοντά στον τοπικό πληθυσμό, Ε, κάνει κάποιο λαθρομπόριο, κάποια δικής, αλλά έχει και ε, κάποιες αρχές, κάποιες πεπιθήσεις. Δεν είναι πάντως τόσο συστηματικά οργανωμένες αυτές ε, οι ομάδες. Μεταξύ τους είναι οργανωμένες οι ομάδες, έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Οι σχέσεις τους όμως είναι ρευστές οι σχέσεις μεταξύ τους. Υπάρχουν ε, διαιρέσεις, ε, χωρίζονται, ξαναβρίσκονται ανάλογα με τους ηγέτες τους και... Πολλές φορές δεν μπορούμε να έχουμε επαφή και εικόνα για όλους αυτούς. Τώρα η, τρο... η αντιμετώπιση τρομοκρατίας ε, είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών, η αστυνομία, και πολλοί άλλοι φορείς και βέβαια το προληπτικό σκέλος είναι σημαντικό. Έχουμε και ένα σκληρό πύρινα εξτρεμιστών σε πολλές συνιστώσεις, αλλά κάποιοι άλλοι πηγαίνουν σε κάποια τέτοια ομάδα γιατί τους υποσχέθηκαν χρήματα. ή ε, τους είπαν κάποια πράγματα. Όλες αυτές οι ε, καταστάσεις είναι ρευστές και δύσκολες. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούμαστε με την πρόληψη της ρίζοσπαστικοποίησης και την αποτροπή της τρομοκρατίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορούμε να αποτρέψουμε, να προλάβουμε μια επίθεση, φυσικά και αυτό είναι πάρα πολύ καλύτερο, δεν είναι εύκολο βέβαια. Την πρόκληση πάντως την έχουμε δεχθεί και πρέπει ε, να ελέγξουμε και να κατανοήσουμε τους διάβλους μέσα από τους οποίους περνάνε όλα αυτά. Υπάρχει η ομάδα εργασίας OS Έχουμε σχέση με τις αντιπροσωπείες. Η Μαυριτανία εργάζεται στενά σε συνεργασία με, σε συνεργασία με εμάς. Οι θρασκευτικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις προσπαθούν να πείσουν γιατί πολλοί που ε, δραστηριοποιούνται μέσα σε μια τρομοκρατική ομάδα δεν έχουν πλήρη επίγνωση του τι κάνουν και πρέπει λοιπόν να, το, να τους ε, βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση τον κύριο Μπράιαν, τον ειδικό απεσταλμένο, χαίρομαι πάντα όταν τον συναντώ. Δεν έχουμε συχνές επαφές, αλλά είχαμε προβλέψει να πάμε μαζί στη Λιβύη. Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Πάντως είναι παρόν και είναι καλό όλοι να είναι παρόντες. Τώρα αν είναι καλύτερα συντονισμένοι τρομοκρατές από τη διεθνή κοινότητα λιγότερο, είναι ολιγάριθμοι, πιο ολιγάριθμοι από σε σχέση με εμάς και έχουν λιγότερα μέσα ε, στην ε, διάθεσή τους. Όμως δεν είναι και τελείως λάθος ότι μπορεί να είναι πιο καλά συντονισμένοι. Έχουμε και όλη αυτή την κλίμακα Σαχάρα Σαχέλ, έχουμε την Ποσαχάριο ε, Αφρική, τη Βόρεια Αφρική, τις δύο αυτές διευθύνσεις επειδή υπάρχουν αυτέ οι δύο διευθύνσει και υπάρχει πρόβλημα συντονισμού, ναι, αποκτούν ένα πλεονέκτημα μέσα σε αυτέ τι τρομοκρατικέ ομάδε, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ε, το κατανοούμε και αρχίζουμε να δουλεύουμε καλύτερα. Υπάρχει όμω κινητικότητα των τρομοκρατικών ομάδων και αυτό είναι ένα θέμα. Το Μουζάου επίσης βλέπουμε ότι προχωράει εκεί που στρατολογούσε ε, πολύ έτσι ε, ντόπιου κυρίω, τώρα στρέφεται και προς τη Λιβύη και στο αστικό, στα αστικά κέντρα, για τη Συρία για παράδειγμα ισχύει αυτό που λέω, ε, εκεί μπορεί κάθε να βρίσκει πιο ενθουσιώδη σε σχέση με την επαρχία. Υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, διστακτικές κινήσεις που γίνονται σιγά σιγά. Η Λιβύη είναι το βασικό θέμα. Δεν έχουμε ακόμη βρει τα κλειδιά για να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα, για τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ εγώ βέβαια να κρίνω τα κράτη-μέλη, αλλά είμαι προσιλωμένο στο στόχο να προωθήσουμε μια κοινή δουλειά για τα Σαχέλ, να δημιουργήσουμε δηλαδή ε, ε, έτσι, μια, ένα πλαίσιο καλύτερου συντονισμού. Έχουμε συναντηθεί μια φορά στην Ισπανία, θα συναντηθούμε στη Γερμανία θα πρέπει όλοι αυτοί που παρακολουθούν τα θέματα του Σαχέλ να μπορούν να συναντώνται, να συνεργάζονται. Δεν είναι ε, μια από τις μας ίσως, δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά πρέπει ίσω και να βγούμε από το αυστηρά τυπικό και επίσημο πλαίσιο. Εγώ έχω εργαστεί σε πολλά κράτη-μέλη και έχω πει ότι ναι, εγώ μπορώ να επισκεφθώ όλα τα κράτη-μέλη για να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να παγιώσουμε αυτό το κοινό όραμα, να καταλάβουμε τις προκλήσεις, τι διακυβεύεται, να έχουμε μια κοινή βούληση σταθερή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι λείπει πιο πολύ. Ε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και πρέπει να το αναζητήσουμε, πιστεύω, σε αυτό το κοινό όραμα, το πραγματικά εναρμονισμένο όραμα. Η σχέση με τη ΣΥΠΑ. Έχουμε πολύ συχνές επαφές σε πολλά επίπεδα και φόρα. Έχω πάει και εγώ στην Ουάσιγκτον και έχω συναντηθεί με τους αρμόδιους εκεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι ε, πιο πολύ εδώ και δέκα χρόνια ε, στο τεχνικό και στρατιωτικό σκέλος πιο πολύ δραστήριες ε, και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στις πληροφορίες που παρέχουν έχουν επαφέ με πολλέ χώρε, οργανώνουν κοινέ στρατιωτικέ ασκήσει με πολλέ χώρε. Έχουμε πολύ καλή σχέση και πολύ καλό διάλογο γιατί έχουν στρατηγικό όραμα και έποψη για την ε, περιοχή την ευρύτερη. Και οι ΙΠΑ ε, έχουν την τάση να θεωρούν ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλη πρόκληση ε, για την ασφάλεια Βόρεια Αφρική Σαχέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασχοληθεί, λένε οι ΙΠΑ, πιο στενά παρέχουν επίσης, ε, μάλλον προσφέρουν πολύ συγκεκριμένες τεχνικές υπηρεσίες. Και σε επίπεδο πρεσβειών και επίπεδο άσκητων μας λένε θέλουμε να σας βοηθήσουμε, μπορούμε να σας ε, βοηθήσουμε. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν πολύ, είναι πολύ δικτυωμένοι και δραστήριοι στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν θέλουν να έχουν ηγετικό ρόλο για πολλούς λόγους, πολιτικούς τα κτλ. Όμως είναι δετεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν φαντάζομαι ότι τα κάλυψα όλα, αλλά αρκεί μάλλον έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη. Πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας ξαναέχουμε εδώ, να σας ξανακούσουμε. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ και πολύ καιρό και που θα συνεχίσει να μας απασχολεί πέρα από την επικαιρότητα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η αποστολή σας είναι δύσκολη, περίπλοκη και ελπίζουμε τα αποτελέσματα να μην αργήσουν και να είναι πολύ θετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα μας, τον κύριο Σεράνο. Καλό τον κύριο Ποπόφσκι, τους επόμενους ah, Bonjour.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 Bien, chers Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι όσοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τη συζήτηση για το Σαχέλ μπορείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα γιατί εμείς περνάμε στο δεύτερο θέμα που είναι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Εν μέρη το Συμβούλιο αυτό είχε σαν θέμα την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ο καθένας ε, μπορεί να παρουσιάσει τα δικά σου συμπεράσματα, προσωπικά και πολιτικά. Εγώ τουλάχιστον απογοητεύτηκα από τα αποτελέσματα αυτά. Μάλλον ε, δεν περίμενα και τίποτα, άρα ήμουν σχετικά απογοητευμένος θα έλεγα από το αποτέλεσμα. Λυπούμε παρόλα αυτά που μια τέτοια ευκαιρία, μια συνάντηση κορυφής και με πολύ περιορισμένα βεβαίως ε, αποτελέσματα, δεν μας άφησε παρά μόνο ένα μισοάδιο ποτήρι. Κάποιοι άλλοι ίσως βέβαια είδαν το ίδιο ποτήρι μισογεμάτο, ανακοινώνοντας ένα χρονοδιάγραμμα και κάποια αποτελέσματα. Από την άποψη λοιπόν καθαρά της δικής μας υποεπιτροπής και από αυτά τα οποία εμείς έχουμε παρουσιάσει και ψηφίσει την της έκθεση της κυρίας Κοπά, την έκθεση του κυρίου Γκάλερ, εμείς πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολύ πιο φιλόδοξες προσδοκίες γιατί θεωρούμε ότι η άμυνα είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να είμαστε απολύτως ρεαλιστές. Βεβαίως θα συμφωνήσω με το ρεαλισμό των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, παρόλα αυτά περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια κάτι παραπάνω. Ολοκλήρωσα την ε, εισαγωγή μου, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να υποστηριχθεί από όλους. Είμαστε ακόμα στον Ιανουάριο, αρχή του χρόνου και με τις ευχές για ένα ευτυχισμένο καινούριο χρόνο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σεράνο, ο οποίος είναι σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής ε, του Πρόεδρου του Συμβουλίου, να πάρει το λόγο για να σχολιάσει τα πρώτα θέματα μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας, μια πολιτική με περισσότερο συντονισμό. Κύριε Σεράνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που με προσκαλέσατε και συγκαλέσατε αυτήν την ε, συνεδρίαση που αποδεικνύει την αφοσίωση του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόθεση του όλου θέματος. Όντως η απογοήτευσή σας είναι πραγματική, αλλά θα μας δώσει και την πολιτική όθηση για να προχωρήσουμε, ελπίζω. Δεν είναι μόνο αρνητική, λοιπόν, ως συνέστημα. Στην έκθεση που αναφέρατε αναφέρονται κάποιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αλλά όλα αυτά μας ε, οθούν στο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί θα παραμείνουν ε, σημαντικά και θα αξιοποιηθούν ώστε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Και η διαδικασία αυτή να εξελιχθεί τα ερχόμενα χρόνια ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, θέσουν τον εαυτό τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να αναλάβουν καλύτερα τις ευθύνες τους, τις ευθύνες που τους αναλογούν, για να ε, προσφέρουν ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Και αν δεν σας πειράζει, τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. The, θα ήθελα λοιπόν εδώ να παρουσιάσω τα συμπεράσματά μας στα μέλη της Επιτροπής σας και να ελπίζω στη στήριξή σας στην όλη διαδικασία αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι τα επιτεύγματά μας ως σήμερα. Ξέρετε ότι η διαδικασία ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012 με τα συμπεράσματα ακριβώ του Συμβουλίου με συγκεκριμένη εντολή προ την ΥΠΑΤΗ πρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό τη Άμυνα, για να εργαστούν σε τρει άξονε: Την αποτελεσματικότητα της κοινή πολιτική, την ανάπτυξη των, δυνατοτήτων μας, των μάχημων δυνατοτήτων την ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων. Άμυνα δηλαδή με βιομηχανία βασισμένη στην τεχνολογία στην Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στο ύπατο επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβόλαιο και έτσι το 2013 είχαμε μια πολύ γόνιμη προσπάθεια διότι ακριβώς συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από, την, από τον επιχειρηματικό κόσμο, τους θεωρητικούς και ακαδημαϊκούς, τους εμπειρογνώμονες, το Συμβούλιο, την ΕΕΔ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την, τον Οργανισμό Άμυνας. Όλοι συνεργάστηκαν προτείνοντας ιδέες για να προχωρήσει η πορεία, η διαδικασία. Σημαντικά επιτεύγματα της διαδικασίας αυτής ήταν η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όλοι γνωρίζετε, η έκθεση της ύπατης εκπροσώπου που οδήγησε σε μια πρώτη φάση στην έγκριση ουσιαστικών συμπερασμάτων από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο που αν τα κοιτάξετε αναφέρουν τουλάχιστον 40 διαφορετικές ε, δράσεις που θα πρέπει να αναλυθούν. Επίσης υπάρχει και επικοδομητικός διάλογος αλλά και έγκριση συμπερασμάτων το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο είχαμε πάλι έγκριση συμπερασμάτων με 19 διαφορετικές δράσεις και ε, ακόλουθες δράσεις που θα πρέπει να προωθηθούν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου θα έλεγα, έγινε μια ανεπροηγουμένου συζήτηση που είχε πολλά χρόνια να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Το ζήτημα καλύφθηκε τόσο διεξοδικά που πραγματικά ήταν η πρώτη φορά η συζήτηση ξεκίνησε αμέσως πριν την ε, επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του καθεαυτού και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ε, έκανε μια παρουσίαση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ε, στηρίζοντας την, ε, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως κατά την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας τους και της αμυντικής τεχνολογίας τους, αλλά και των στρατηγικών δυνατοτήτων των κρατών μελών. Αυτό ακολουθήθηκε από μια ενεργό ε, ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των, κρατών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μια συζήτηση που κάτσε πάνω από ένα δύο ώρο, μια πραγματική συζήτηση επί της ουσίας, από την οποία θα μπορούσε κανείς να κρατήσει τέσσερις βασικές ιδέες. Η πρώτη και η πλέον σημαντική ήταν η πραγματική ε, δέσμευση των 100 μελών στην ε, συνειδητοποίηση ότι πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες για να υπάρξει ασφάλεια στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να τα αφήσουν αυτά στις παρελθούσες διευθετήσεις, αυτές που είχαμε γνωρίσει ως σήμερα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται σε άλλη θέση πλέον, οπότε θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές χώρες να βεβαιωθούν ότι έχουν τις δυνατότητες για να αναλάβουν τις ευθύνε τους και να μην ε, αφαιθούν στο κενό που έχει δημιουργηθεί, διακυβεύοντας την ε, ασφάλεια την δική μας και των γειτόνων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Έπειτα, από αυτό το συμπέρασμα προέκυψαν άλλα. Δηλαδή, τι ε, εξυπακούει η ιδέα αυτή. Το βασικό στοιχείο στις συζητήσεις είναι ότι χρειάζονται απαραίτητες αισθητικές ε, δυνατότητες, τις οποίες δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και έχουν αλλάξει. Είναι διαφορετικό το περιβάλλον μας, ε, διαφορετικές εκθέσεις και αναθεωρήσεις έχουν ετοιμαστεί, υπάρχουν νέα όπλα και γι' αυτό και εμείς χρειαζόμαστε νέα μέτρα για να απαντήσουμε, να αποκριθούμε στις διάφορες ανάγκες. Για τις δυνατότητές μας η αμυντική βιομηχανία θα πρέπει ακριβώς να υποστηρίζει αυτές τι τις δυνατότητες, το ίδιο και η τεχνολογική βάση που απαιτείται για την αμυντική βιομηχανία. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα των αρχηγών και των κυβερνήσεων στις συζητήσεις τους. Ένα άλλο σημείο που το τόνισαν επίσης πολύ τότε ήταν η συνολική προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι δεν μπορεί κανείς να καλύπτει μόνο με στρατιωτικά μέσα τις ανάγκες της ασφάλειας, αλλά χρειάζεται μια ποικιλία από εργαλεία. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώ το σημείο που μπορούν να συναρθρωθούν σωστά όλα αυτά τα εργαλεία για να είναι αποτελεσματικά. Θα πρέπει όμω να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και να είμαστε συνολική ε, στην προσέγγιση μας, ε, να ακολουθήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Όχι μόνο για τη διαχείριση των κρίσεων που αφορούν τους πολίτες, αλλά για θέματα πολιτικής που μπορεί να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων. Θέματα που επίσης τονίστηκαν από πολλούς ε, αρχηγούς και κυβερνήσεων που πήραν τον λόγο. Το άλλο σημείο όπου οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πολλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνη. Πρέπει να συνεργαστεί με του διεθνεί εταίρου τη και υπάρχουν πολλοί στρατηγικοί εταίροι και οργανισμοί με του οποίου μπορούμε να συνεργαστούμε, όχι μόνο το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ φυσικά πρωτίστω, αλλά υπάρχει ο ΙΕ, η Αφρικανική Ένωση και άλλοι. Ακόμα και στην Ευρώπη έχουμε τον, ΟΑΣΕ, καθώς και άλλε άλλες χώρες εταίρους. Όταν λοιπόν επεμβαίνουμε και κάποιες φορές μακριά από τα σύνορά μας, σκέφτομαι τώρα τη δική σας παρουσίαση, την παρουσίαση που ακούσαμε πριν από την δική μας, όταν λοιπόν σκέφτεται κανείς τέτοιες περιπτώσεις, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχει επέμβαση, αλλά να μπορούμε και να βοηθήσουμε τα κράτη στα οποία δρούμε, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες και να έχουν την δική τους ασφάλεια. Αυτό δεν ήταν μόνο μέρο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, αλλά και των μηνυμάτων που ήθελαν να τονιστούν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων. Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα ήταν η συμπληρωματικότητα και η ανάγκη συντονισμού και καλή ε, αγαστή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Η παρουσίαση βεβαίω του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ήταν ακόμη πιο σαφή ω προ το σημείο αυτό, αλλά ήδη έχουμε θετικέ εμπειρίε από τη συνεργασία μα και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί. Το τόνισαν οι περισσότεροι από όσου πήραν το λόγο. Τέλο, η σημασία μια αυξημένη και εντατικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων ε, και εμπλεκόμενων φορέων, Κύρίω των κρατών μελών. Αυτό το σημείο τονίστηκε όλος ιδιαίτερο όταν μιλήσαμε για την ανάπτυξη των αμυντικών μα δυνατοτήτων, όχι μόνο για την ανάπτυξή του αυτή καθεαυτή, αλλά και για την ε, λειτουργία του και για την συντήρησή του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδου τη συνεργασία και το οποίο το ανέφεραν πολλοί τότε, είναι Νομίζω το, ε, το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου της ε, αεροπορικής, της ελληνικής αεροπορίας. Ε, εδώ νομίζω ότι όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, τα αεροπλοϊκά μας μέσα, ώστε να τα συνδυάσουμε και να έχουμε άμεση απόκριση όπου χρειάζεται. Τώρα, ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε τώρα. Η βασικότερη πρόκληση είναι η υλοποίηση όλων αυτών των αποφάσεων και μια από τι πρώτε δυσκολίε είναι να διατηρήσουμε το ρυθμό ε, υλοποίηση που είχαμε και το 2013. Αυτή είναι μια πρώτη σίγουρα μεγάλη πρόκληση και εδώ το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει καθιεραστικό ρόλο. Μπορεί να μα βοηθήσει το ρυθμό αυτό να το διατηρήσουμε αμύωτο. Νομίζω η συνάντηση αυτή είναι μια πρώτη απόδειξη αυτή τη πρόθεση. Το επόμενο ραντεβού ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2015, οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν εντωμεταξύ υλοποιήσει τις δράσεις που αναφέραμε μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Κάποιες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2014 και μάλιστα είπατε εκπρόσωπος εμ, δέχτηκε την έκκληση να ετοιμάσει ε, έκθεση μέσα στο 2014 που να είναι έτοιμη για την επόμενη χρονιά. Είναι προφανές ότι το να διασφαλίσουμε το να υπάρχει ασφάλεια, το να έχουμε τις δυνατότητες που χρειαζόμαστε, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε ένα, δυο ή τρία χρόνια. Τρόπον την άλλη λοιπόν θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις ε, για τις οποίες όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Πρέπει να έχουμε όλοι αυτό το στόχο υπόψη μας και έχουμε εντοπίσει τομείς όπου μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες όπως τα εξαποστάσεως ε, τηλεχειριζόμενα αεροπορικά συστήματα, οι δορυφόροι, ε, οι δορυφόροι ε, και άλλα σημεία της όλης διαδικασίας που θα εντοπιστούν στη συνέχεια. Για το σκοπό αυτό έχουν οργανωθεί αρκετέ ε, συναντήσει, νομίζω όμω θα μα τα αναλύσει καλύτερα ο Μάτζεκ Ποπόφσκι. Ε, μια σημαντική διάσκεψη που έχει προβλέψει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα το Μάρτιο για να μπορέσουμε να ξαναδούμε με λεπτομέρειε τα θέματα αυτά, να τα προωθήσουμε. Επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει διάσκεψη με όλου του ενδιαφερομένου στι 4 Μαρτίου. Διάσκεψη που θα ορίσει μια σειρά προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία για να συνεχίσει να συνεισφέρει από τον τομέα των αρμοδιοτήτων της. Θα υπάρξουν υπουργικέ συναντήσεις. Νομίζω ότι ο Μάτζεκ Ποπόφσκι θα εξηγήσει πώς η διαδικασία αυτή μπορεί να προχωρήσει με την ενεργό συμμετοχή και τις συμβολές που προβλέπεται να έχουμε. Από την πλευρά μας θα φροντίσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει και συνέχεια και ενθάρρυνση θα κοιτάζουμε μεγάλη προσοχή πώς στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που ήδη έχουν προγραμματιστεί μπορούμε να έχουμε συνέχεια της διαδικασίας και να ενθαρρύνουμε καθώς προχωρούν τα πράγματα να συνεχίζεται. Κάποιες σύνοδοι έχουν ήδη προβλεφθεί. Έχουμε μια κοινή συνοδοκορφή με την Αφρικανική Ένωση, μεγάλους ε, σημαντικούς εταίρους μας που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ενέργειές μας και θα δούμε εάν μπορεί να προκύψουν συμπεράσματα και από αυτή τη συνάντηση για να χρηματοδοτήσουμε λόγω χάρη τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση. Σημαντικά στοιχεία των συμπερασμάτων. Πώς μπορούμε καλύτερα να εξοπλίσουμε και να εκπαιδεύσουμε τις χώρες που βοηθούμε. Επίσης άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του Αφρικ... της αφρικανικής ε, δύναμης έγκαιρης αντίδρασης. Αυτά θα τα δούμε στη Σύνοδο Κορυφής με την Αφρική. Και στο σκηνικό του αφρικανικού αρχιτεκτονήματος για την ασφάλεια και την άμυνα. Υπάρχει και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο, πολύ σημαντική και αυτή, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρουσιάσει το έργο που έχει προβλέψει και επιτελέσει ως τότε, κυρίως ως προς τις πρόσθετες δυνατότητες, τις μα μας δυνατότητες, που θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και Υπάρχουν και κάποιες διμερεί, διμερείς ε, συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι πια μυστικό ότι θα έχουμε μια σύνοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ομπάμα θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής. Νομίζω ότι είναι η πρώτη επίσημη επισκεψή του στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη Μαρτίου. Οπότε θα έχουμε και πάλι μια ευκαιρία να ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα και να παρουσιάσουμε το έργο που φέρνουμε εις πέρας προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ σημαντικός στο να για να προχωρεί αυτή τη διαδικασία, επειδή ακριβώ συζητήθηκαν όλα αυτά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και επειδή προσπαθούμε να συντονίσουμε του διαφορετικού φορεί οι οποίοι συνεργάστηκαν σε ένα κλίμα αρμονικό. Ε, πράγμα το οποίο είναι όντω αξιέπαινο και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θα συνεχίσει το έργο του στην στήριξη όλη αυτή τη διαδικασία που θα θέλαμε να προχωρήσει ομαλά. Ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο που μου δώσατε για την ομιλία αυτή. Είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, Εγώ πραγματικά πάντα θεωρούσα τον κύριο Σεράνο σαν ένα εξαιρετικό Ευρωπαίο διπλωμάτη. Μου επιβεβαιώνεται αυτή την εντύπωση. Και με πείσατε πραγματικά όσον αφορά το ρόλο που θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκώντας πίεση για όλη αυτή τη διαδικασία. Η παρουσίασή σας ήταν ε, πλήρης, ενδιαφέρουσα. Εκεί που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι σε αυτό που είπατε όσον αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου. όσον αφορά την ε, ουσία αυτών των συζητήσεων, τη συνοχή και πραγματικά είναι πρώτη φορά από το 2008 που πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Κύριε Ποπόφσκι, από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ήμουν λίγο επικριτικός στην ε, εισαγωγή που έκανα όσον αφορά την υπατή εκπρόσωπο. Η έκθεση που μας παρουσιάσατε ήταν πολύ ουσιαστική και περιείχε πολλά στοιχεία για το ρόλο του Κοινοβουλίου και για τις προσπάθειες συντονισμού. Τι έχετε να πείτε μετά το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πραγματικά ήθελα να πω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να εντοπίσει πολλά μηνύματα, ίσως όχι στα συμπεράσματα, αλλά στο κείμενο της έκθεσης ε, της ε, ΕΠΕ της Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα πολυθετικά σας σχόλια. Συνοπτικά, αν ήθελα να πω με μια φράση τι έγινε το Δεκέμβριο, θα έλεγα ότι οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η άμυνα είναι αυτό που έλεγε ο Helmut Kohl, υπόθεση των αρχηγών, των επικεφαλής. Έβαλαν λοιπόν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, αποφάσισαν να το διατηρήσουν και αυτό βεβαίω επιβεβαιώθηκε σαν γεγονό. Το 2013 ήταν ένα έτος μεγάλης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, δηλαδή προετοιμάσαμε αυτό το Συμβούλιο η ανακοίνωση ότι θα συζητηθεί το θέμα σίγουρα δημιούργησε μια πολιτική κίνηση, όθηση και πολύ όχι μόνο στον θεωρητικό και ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και από τον βιομηχανικό κλάδο των εξοπλισμών, στήριξαν αυτή την κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν γιατί και εσείς υποστήριξατε αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιανουάριο του 2013 θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα θετικό αποτέλεσμα όλων αυτών θα ήταν αν οι ηγέτες δεσμευθούν, αν υπάρξουν προτάσεις για κάποια προγράμματα συνεργασίας και βεβαίως να υπάρξει έκφραση δέσμευσης από μέρους των Ευρωπαίων ηγετών. Και όλα αυτά τα πετύχαμε. Και βεβαίως ξεκίνησε η συνάντηση και μάλιστα τα συμπεράσματα αυτού του Συμβουλίου με τη φράση ότι η άμυνα και η ασφάλεια είναι κάτι που σημαίνουν πολλά για την Ευρώπη. Αυτό είναι μια δυναμική φράση που τα λέει όλα ουσιαστικά. Τα κράτη-μέλη ζητούν πιο ουσιαστική στρατηγική συζήτηση και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο μέλλον σε μία αλλαγή του στρατηγικού περιβάλλοντος. Δεν λέω ότι θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί την διατύπωση μιας νέας στρατηγικής, αλλά μία από τις προτάσεις είναι και αυτή και ξεκινάει η διαδικασία. Πιστεύω λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η νέα κατεύθυνση, η νέα στρατηγική. Ακούσαμε πολλά επικριτικά σχόλια, αλλά και κάποια θετικά. Και αυτό εκτός Βρυξελών. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο από θεωρητικούς και καθηγητές, αλλά και από ανθρώπους ε, ειδικού στον κλάδο, που συνήθως ήταν αρνητικοί κάθε φορά που ξεκινούσε μια προσπάθεια να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της και της άμυνας. Σήμερα λοιπόν για τα επόμενα δύο χρόνια έχουμε καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει η γενική κατεύθυνση της μελλοντικής μας εργασίας και συμπεράσματα από το Συμβούλιο που μας δίνουν διάφορες ιδέες, κατευθύνσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας με κάποια προγράμματα που βρίσκονται το καθένα σε διαφορετικό βαθμό οριμότητας και εξέλιξης και θα αναφερθώ εδώ στη στρατηγική για την θαλάσσια ασφάλεια που θα υιοθετηθεί τον Ιούνιο του 2014. Η απόφαση λήφθη τη Δευτέρα όσον αφορά την προετοιμασία του σχεδιασμού για μία αποστολή για την Κεντρική Αφρική. Η εντολή έχει δοθεί ήδη στην Ιβαντή εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορώ να επανέλθω στο θέμα αυτό αν σας ενδιαφέρει απαντώντας στις ερωτήσεις σας. Πριν τον Ιούνιο του 2015 υπάρχουν βεβαίως και πολλές άλλες δυνατότητες να υπάρξει δέσμευση σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Στην Αφρική όπου πολλά από αυτά που καλούμαστε να διεκπαιρεώσουμε συμβαίνουν στην Αφρική. Το πρόγραμμα Train and Equip για κατάρτιση και εξοπλισμό που ισχύει κυρίως για την Αφρική. Τώρα, εδώ στην ίδια πόλη, στο ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αποτελούν πολύ σημαντικά ορόσημα για αυτόν τον οργανισμό. Και βεβαίως η συνάντηση κορυφής του Σικάγο ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργούμε λοιπόν παράλληλα και πραγματικά η άμυνα έχει πλέον γίνει ένα από τα θέματα που σημαδεύουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην περιοχή της Σαχάρας και του Σαχέλ. Συζητήσατε το θέμα αυτό ακριβώς πριν ξεκινήσει αυτή η ακρόαση. Το θέμα των αποστολών αλλά και της ε, χρηματοδότησής τους. Σήμερα περιμένουμε πολλά για τις ε, ενεξελίξει αποστολές στην Αφρική και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί αυτές οι αποστολές να αποκτήσουν λίγο περισσότερη ευελιξία. Επίσης, μια συστημική θα λέγαμε ανάθεση όσον αφορά τα προγράμματα μακροχρόνια στρατηγικής συνεργασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξουν επικαλύψεις στον σχεδιασμό και να μην υπάρχουν γενικότερα επικαλύψεις με τον ΝΑΤΟ. Βεβαίως και θα συνεργαστούμε εδώ σε πολύ εντατικούς ρυθμούς με τα κράτη-μέλη, με τους αρμόδιους υπουργούς. Θα συνεργαστούμε σε στενά και με την Επιτροπή για θέματα βιομηχανίας εξοπλισμών. Όμως πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ φορτωμένο χρονοδιάγραμμα αυτό των δύο επόμενων ετών. Η στόχοι μας είναι σαφής. Είμαστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι πρόκειται για κάτι το πολύ ενθαρρυντικό που μας ε, στηρίζει και βεβαίως συνεργαζόμαστε και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς πέρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci. On Ευχαριστώ πολύ. Ας ε, κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το πρώτο κομμάτι. Τρεις έχουν στήσει λόγο. Πρώτος ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές Νομίζω ότι οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτά που θα μπορούσαν να μην συμβούν καθόλου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι κάπου στη μέση. Μπορεί κανείς να εργαστεί περαιτέρω, μπορεί κανείς να περιοριστεί σε αυτά τα συμπεράσματα, μπορεί να παραμείνει σε αυτό και να περιμένει κάποιες επιπλέον προτάσεις της Επιτροπής. Όλα μαζί όμως, κατά κάποιο τρόπο, μας δημιουργούν μια ουσία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μια βάση και έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα αυτή είναι και η άμεση γειτονιά μας, η πολύ κοντινή μας γειτονιά, η Αφρική, η Κεντρική Αφρική μας δείχνουν σήμερα ότι οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να είναι πανταχού παρόντες και είμαστε υποχρεωμένοι να επέμβουμε. Δεν μπορούμε διαρκώς να περιμένουμε τους εταίρους μας από την Αμερική να αναλάβουν το βάρος αυτών των αποστολών. Και θεωρώ πραγματικά ότι η αναθεώρηση του μηχανισμού Αθηνά είναι κάτι που θα πρέπει να μας αποσχολήσει. Εδώ στην Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δυνατότητες, ότι χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό χρηματοδότησης που να λειτουργεί και να μπορούμε να τον επικαλεστούμε και σε κάθε περίπτωση πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα σωστό ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην Ευρώπη. Και εγώ πάντα θυμάμαι αυτό που είχε πει η Άννα Στην Πορτογαλία έχουμε δυνατότητες, έχουμε ενόπλες δυνάμεις. Αλλά δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να αναλάβει μόνη της σήμερα μια τέτοια αποστολή. Ο καθένας έχει τις δικές τους δυνατότητες, τις οποίες προσπαθεί να αναπτύξει, αλλά ο καθένας από εμά μόνος του δεν μπορεί και δεν πρέπει να ε, κάνει καμία τέτοιου είδους αποστολή. Χρειάζεται λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένας μηχανισμός καινούριο, αναθεωρημένος και αυτό θα είναι και η δυνατότητα να συνεισφέρουμε όλοι σε τέτοιες αποστολές. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλες αυτές οι πτυχές που μας παρουσιάσατε που αφορούν τα δύο επόμενα χρόνια, το χρονοδιάγραμμα, τους στόχους, τη χρηματοδότηση, τον εξυγχρονισμό. Είναι πολύ φιλόδοξη στόχη και είμαι σίγουρος ότι ναι, ο χρόνος μας πιέζει μέχρι τα μέσα του 2015 και σίγουρα ακόμα και αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2015 θα έχουμε πετύχει πολλά. Ελπίζω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα αυτό της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης, θα εκτελέσουν αυτό το έργο με αποτελεσματικότητα. Βλέπω ότι έχουμε ξεκινήσει στη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα. Και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να υλοποιηθούν και στην πράξη αυτά που σήμερα έχουμε εκφράσει. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Ε, Νομίζω Βεβαίως καταλαβαίνω ότι η δουλειά σας είναι να μας παρουσιάσετε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό την καλύτερη οπτική γωνία τα πράγματα που σας αφορούν. Αλλά παρά τις προσπάθειές σας δεν καταφέρω να πιστέψω το Συμβούλιο πιστεύει στα ζητήματα άμυνας. Είναι σαν την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Στα λόγια και στη ρητορία βλέπουμε πάρα πολλά, αλλά στην πράξη τίποτα δεν γίνεται. Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Μάλλον το αντίθετο. Βλέπουμε να ανακοινώνεται γενοκτονία στην κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και οι υπουργοί μας να αποφασίζουν μια κλασική αποστόλη ασφάλειας και άμυνας που θα πάρει εβδομάδες να ε, κινητοποιηθεί. Ενώ θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους μάχημους χρηματισμού που ήδη διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβουν δράση. Και ξέρω ότι με τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό η Γερμανία θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω για την Ευρωπαϊκή Άμυνα Αναγνωρίστηκε όμως, ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η επιχείρηση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία είναι μια σημαντική κίνηση, αλλά όλοι μας λένε δεν θα συμμετάσχουμε. Ε, περίμενε κανείς να υπάρχει άλλο είδος στήριξη για αυτή την επιχείρηση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε τι καταλαβαίνουμε, ότι κανείς δεν το αντιλαμβάνεται αυτό σαν να μας αφορά άμεσα το θέμα. Και με συγχωρείτε κύριε Παπόφσκη, αλλά τι μας λέτε ότι στο θέμα αναθεώρησης της δημοσιονομικής κατανομής του κόστους θα πάμε στις Βρυξέλλες να το, θεωρήσουμε. Εγώ αυτό νόμιζα θα κάνει η περασμένη σύνοδος. Ένα χρόνο τα συζητάμε τα λέμε και τα ξαναλέμε. Το Ευρωκοινοβούλιο έκανε τη δουλειά του. Έκανε αυτό που έπρεπε. Τι συνεισφορέ του, όλη την πολιτική στηρίξη τα προσέφερε στο Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα. Και μα λέει, καλά, καλά, θα το κάνουμε σε μερικά χρόνια, περιμένετε λίγο. Δεν γίνεται τίποτα εντωμεταξύ. Και επήγει το θέμα. Φάνηκε αυτό από την EUCAR, ε, την, αυτή την αποστολή και να σας πω και κάτι άλλο, ε, Κούκου, τι γίνεται με την ε, θαλάσσια ασφάλεια. Δεν θα γινόταν μια σύνοδος αυτό, ε, για το θέμα αυτό, για την ασφάλεια στη θάλασσα. Εμείς τη δουλειά μας δεν κάναμε. Το Συμβούλιο τι έκανε και πώς μεταφράζεται αυτό σε πράξη. Για πείτε μας. Ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι συντονισμός υπάρχει μεταξύ ή έστω ε, ανατίθεται από την είπατε εκπρόσωπο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ που είναι άσχετα μεταξύ τους και έχουν να κάνουν με τη δράση στη θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την DG Mare, την DG Move, την DG Home και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάνει τίποτα Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ε, θαλάσσια ασφάλεια και άμυνα. Θα περιμένω την επόμενη, τον επόμενο γύρο για να μιλήσω για τι δυνατότητε, τις δυνατότητες και την βιομηχανία μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Φανόρντεν, ο οποίος υποψιάζομαι ότι θεώρησε την σύνοδο αυτή τεράστια επιτυχία. Πρόεδρε, νομίζω όλοι μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά μας στο Συμβούλιο Άμυνας. Πάνω απ' όλα πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Σεράνο και τον κύριο Ποπόφσκι που μας παρουσίασαν όλα αυτά τα στοιχεία εδώ. Νομίζω μπορεί να πει κανεί με ασφάλεια ότι το Συμβούλιο Ασφάλειας ήταν απογοητευτικό. Το Συμβούλιο Άμυνα, μάλλον, ήταν απογοητευτικό. Το περιμέναμε όλο το χρόνο. Περιμέναμε να απογειωθεί η ενία πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Και τι έγινε. Ελάχιστα πράγματα. Ψίχουλα μας δώσανε. Είναι η τρίτη φορά σήμερα που ακούω τον αριθμό των 49 ε, σημείων που θα πρέπει να βιλοποιηθούν και το ραντεβού για το 2015. Εντάξει. Και εγώ θα ήθελα, εάν γίνεται για να μην ψάχνουν οι βοηθοί μου στα τυφλά, να μου δώσετε ένα κατάλογο με τα 49 αυτά σημεία. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερος και ένα-δυο ακόμη σχόλια. σε παρένθεση πάντοτε, στο περιθώριο των όσων λέμε. Δεν είχε τίποτε το μοναδικό, ούτε το καινοτόμο η ενιαία αυτή προσεγγίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έκαθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθούσε να κάνει. Να προσετεριστεί αυτήν την ιδέα ακριβώς της ενιαίας δράσης. Ακόμη και το ΝΑΤΟ και η δράση μας στο Αφγανιστάν, οι ομάδες ανοικοδόμησης, όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία που θα έπρεπε να υποστηρίζουν τη στρατηγική μας επέμβαση εκεί. Τέτοιες αποδείξεις συνολικής προσέγγισης είναι. Δεν είναι κάτι που είναι φοβερά πρωτότυπο. Αυτό κάνει και το κάθε έθνος ή κράτος όταν ε, παίρνει μέρος σε στρατιωτική επιχείρηση. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν παίρνουν μια κλασική ιδέα και μετά τη μετατρέπουν σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Το παράδειγμά σας. Η εντολή, οι εντολές σε επίπεδο ε, αεροπορικών μεταφορών. Ωραία αυτό υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το περιγράφεται, είναι σαν να είναι κανένα φοβερό παράδειγμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάτε για τις απαρχές. Πηγαίνει πίσω στην πρωτοβουλία για την ίδια άμυνα το 1995. Με συγχωρείτε. Αυτό που ιδιαίτερος με ενδιαφέρει, με συγχωρείτε. Ναι, θα σε, θα ξανα, Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή περιμένουμε στο μευτήριο το δεύτερο εγγόνι μου. Θα σας τα πω εντός ολίγου. Εάν όλα πάνε καλά θα σας ενημερώσω. Για την ε, αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Τι ξέρουμε Ποιος θα έχει την ευθύνη για την ε, εντολή. Η Γιουρέσα θα τα αναλάβει από την ε, Ελλάδα. Ή ποιος θα έχει την ε, εικονική ευθύνη, την ενδιάμεση ευθύνη Πώς θα εκτυπλωθεί αυτή η αποστολή, τι ελικόπτερα θα αποσταλούν, τι αριθμός και τι, πώς, πώς θα υποστηριχθεί οικονομικά αυτή η ενέργεια. Τζέφρι, αύριο το πρωί έχουμε ειδική συζήτηση για την αποστολή της CSDP στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Λοιπόν, ίσως να μην το καλύψουμε τώρα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Παναγιώτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω με βάση τα συμπεράσματα και τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα, έχοντα υπόψη μα ε, τι συστάσει του Συμβουλίου για την ανάπτυξη και την ε, συγκέντρωση των ε, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μέλων, θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό στο άμεσο μέλλον, με δεδομένου του δημοσιονομικού περιορισμού των χωρών μελών. Δεύτερο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε την απόφαση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική Ασφάλεια ή για μια επικαιροποιημένη στρατηγική. Και ταυτόχρονα κάλεσε την είπατε να ε, αξιολογήσει μέχρι το 2015 τις προκλήσεις του στρατηγικού περιβάλλοντος. Ο κύριος Ποπόφσκι ήδη έχει εκφράσει την ε, προθυμία του να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε συνέχεια αυτής της ε, αξιολόγησης θα είναι η χάρεξη μιας νέας στρατηγικής ασφάλειας ή μια επικαιροποιημένη εκδοχή της στρατηγικής αυτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Thank you. Um, uh, just two, three questions. Ακούστηκαν ερωτήματα, αλλά να απαντήσω και σε σχόλια. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω με τη χρηματοδότηση. Το μηχανισμό των Αθηνών, Αθήνα Mechanism, που ούτως ή άλλως θα αναθεωρηθεί. Προβλέπεται ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρησή του μέχρι τα τέλη του έτους. Αλλά πρέπει να επιταχύνουμε λόγω των ε, καθηκόντων που πρέπει να οργανώσουμε και να φέρουμε σε πέρας. Ε, ένα από τα κεντρικά, ίσως το κεντρικό ζήτημα, είναι ο ορισμός του κοινού κόστους. Δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί από τότε που δημιουργήθηκε ο μηχανισμός ε, Αθήνα, το μείζον ζήτημα ήταν πώς ορίζουμε το κοινό κόστος. Αν ε, μπορέσουμε να διευρύνουμε τον ορισμό, αυτό σημαίνει ότι πολλές ανησυχίες των κρατών μελών θα ληφθούν υπόψη, όπως αυτά που είπε η κυρία Γκόμες, για παράδειγμα. Χθε όλοι είμαστε σε αυτή τη συνάντηση που ανέφερε. Πρέπει να το προσπαθήσουμε. Όχι ότι δεν το έχουμε ξαναπροσπαθήσει. Είχαμε πολύ ζωντανή συζήτηση για τη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα το 2011 που είχαμε την προηγούμενη αξιολόγηση του Μηχανισμού Αθήνα και προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το θέμα αυτό με την ε, πιθανή δημιουργία ενός ε, ταμείου, ε, startup fund και τα κράτη-μέλη τελικά δεν έδειξαν προθυμία για κάτι τέτοιο. Εμείς πολλές φορές το προτείναμε, είχαμε διάφορους γύρους συζητήσεων από αυτού δεν το καταφέραμε, αλλά είμαστε υπομονετικοί, θα το ξαναπροσπαθήσουμε και θα έχουμε δύο ε, παράλληλες ε, εργασίες αναθεώρηση του μηχανισμού Αθήνα, χρηματοδότηση στρατιωτικών ε, αποστολών επιχειρήσεων και το δεύτερο μη στρατιωτικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμεσης. Θέλουμε όμως να είναι πιο ευέλικτοι ο τρόπος με τον οποίο θα πάνουμε τους πόρους. Δεν θα συμφωνήσω και δεν θα σας εκπλήξει αυτό βέβαια, ότι δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε κύριε Γκόμες, ότι δεν γίνεται τίποτε. Διότι η απόφαση ε, να δρομολογηθεί αυτή η αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχει εγκριθεί. Κάτι γίνεται λοιπόν ή θα γίνει τέλο πάντων. Και μάλιστα σύντομα. Και τώρα επανέρχομαι. Μάλλον θα επανέλθω σε λίγο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. η συζήτηση για τη θαλάσσια στρατηγική. Δεν είναι κάτι καινούριο, πράγματι. Τώρα όμως έχουμε πολύ καλή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση για μια στρατηγική θα έλεγα ότι σχεδόν επίκειται. Δηλαδή θα προτείνουμε κάποια στοιχεία στρατηγικής αυτής ε, από το Μάρτιο μάλλον ήδη, μέσα στην Άνοιξη δηλαδή, και ελπίζουμε να έχουμε απόφαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Άρα είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Και ο στόχος μας είναι όλοι οι φορείς από κοινού, δηλαδή οι Γενικές Διευθύνσεις Κομισιών και η ΕΔ, για να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Ήδη δηλαδή έχει προχωρήσει το θέμα. Κύριε Βανόρντερ, με τα χαράς, με τα χαράς να σας στείλω τα taskings. Σε όλους, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. σε ό,τι αφορά την ε, γενική αυτή σφαιρική προσέγγιση. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι κάτι καινούριο. Είπαμε απλά ότι θέλουμε να είμαστε πιο συντονισμένοι και πιο αποτελεσματικοί. Έχουμε καλά παραδείγματα και κακά παραδείγματα. Σε κάποιε οργανώσει έχουμε καλύτερο συντονισμό, αλλού όχι. Για τον ΝΑΤΟ πράγματι έχουμε πάρα πολύ καλή ε, εμπειρία με τις ομάδες ανασυγκρότησης ε, επαρχιών, τα PRTs δηλαδή. Τώρα έχουμε συνεργασία με αυτή τη συνολική σφαιρική προσέγγιση. Είναι ένα πλαίσιο πολιτικής, ουσιαστικά ο ορισμός ενός τρόπου σκέψης και δράσης. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα εφεύρουμε κάτι καινούριο. Απλά χρειάζεται βελτίωση του τρόπου εργασίας. Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα έχετε μια ειδική ε, συνεδρία για αυτό το θέμα, αλλά για τις μάχημες ομάδες, τα battle groups, επειδή επανέρχεται το θέμα αυτό και ο πρόεδρος Στρατιωτικής Επιτροπής και το Συμβούλιο στο Συμβούλιο μάλλον έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Η Στρατιωτική Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, η Στρατιωτική Εμπειρογνώμος δηλαδή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μάχημες ομάδες τότε δεν ήταν η προτιμόμενη επιλογή. Πρώτον, διότι υπήρχε περιορισμός ε, στην ανάπτυξη 120 ημέρες και θεωρήσαμε ότι η UFOR ε, για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα έπρεπε να μείνει 4 με 6 μήνες εκεί προς επιβεβαίωση ακόμα. Τώρα, η μάχη με ομάδα η συγκεκριμένη τώρα δεν μπορεί να φέρει σε πέρας όλα, όλες τις στρατιωτικές εργασίες που προβλέπονται. Και δει το συμβουλευτικό ρόλο στην Αφρικανική επιχείρηση Αφίσμα. Και από στρατιωτική πλευράς πρέπει να υπάρχει ομαλή αλληλεπίδραση ε, μεταξύ των επιχειρήσεων της Αφίσμα ε, αλλά και της γαλλικής επιχείρησης. Και επειδή η Γαλλία είναι το κράτος που θα πλαισιώνει αυτή την ε, αποστολή, η Στρατιωτική Επιτροπή κατέληξε ότι είναι καλύτερη επιλογή αυτή παρά να χρησιμοποιηθεί η μάχη με αυτή η ομάδα που έχουμε τώρα. Λεπτομέρειες ε, για το Force Generation και για το ποιος θα είναι ο δικτής δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη. Δηλαδή αυτή τη διαδικασία συγκρότησης των δυνάμεων θα το αποφασίσουμε και περιμένουμε και ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία των Εθνών για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εδώ θα σταματήσω γιατί θα, θα σας πει φαντάζομαι περισσότερα ε, ο συνάδελφός μου στην ε, ειδική συνεδρία που έχετε για την κυρία Παναγιώτοβα. Σε ό,τι αφορά τις μη στρατιωτικές ικανότητες φυσικά έχουμε πρόβλημα και όποτε περιορισμό και όποτε έχουμε μη στρατιωτική ε, επιχείρηση έχουμε ανταγωνισμό με το εθνικό επίπεδο που και εκεί απαιτούνται αυτοί οι πόροι, αυτές οι ικανότητες και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις δυνάμεις όσο το δυνατό. Για το άλλο ερώτημα, ε, ουσιαστικά αυτό που είπα στην εισαγωγή μου. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, μια επικαιροποιημένη μορφή της ή κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε την αξιολόγηση, την εξέταση του στρατηγικού περιεχομένου. Είπατε εκπρόσωπο θα μα κάνει τη σχετική παρουσίαση σε ε, διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και εν συνεχεία το θέμα θα παραπενθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορεί να γίνει κάτι, δεν θέλω να προδικάσω όμως τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι συνεπτική νομίζω η άποψη αυτή, γιατί αν ρωτήσετε τα κράτη-μέλη ατομικά, είναι διαιρεμένα σε σχέση με το κατά πόσο χρειάζεται μια νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση, όχι γιατί είναι κάτι περιττό, αλλά γιατί θεωρούμε όλοι ότι πρέπει πρώτα να γίνει αυτός ο στρατηγικός προβληματισμός και μετά να δούμε τι απόφαση μπορούμε να λάβουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you very much for all the very useful and comment. Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα σχόλια. Πραγματικά εγώ τα ερμηνεύω πραγματικά σε σχέση με τα συμπεράσματα και φυσικά σε σχέση με τη συνέχεια που θα δώσουμε από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμά θέλουν κάτι παραπάνω, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας, σε καμία περίπτωση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως όλοι είπατε, βρισκόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλές από τις δράσεις που πρέπει να αναλυθούν δεν είναι δράσεις που μπορεί να αναλάβει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω οι αφρικανικές χώρες καλούνται εδώ να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο διευκόλυνση, συντονισμού, να χρησιμοποιήσει υπάρχοντες μηχανισμούς, αλλά η ασφάλεια είναι ε, έργο και αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Μόνο ένα κράτος μέλος μπορεί να είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των πολιτών του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια των μηχανισμών της ευρωπαϊκής κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών, μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας, τη μεθοδολογία και σε κάθε περίπτωση εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε βασιζόμενοι στην εμπειρία μας με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε και στα πλαίσια βέβαια της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε δυνατότητες και στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων, αλλά και στην υπόλοιπη δραστηριότητά μας, όπου έχουν γίνει πάρα πάρα πολύ σημαντικοί πρόοδοι αν θέλετε, είμαστε και το μοναδικό φόρουμ εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα αυτά μπορεί να συμβούν σε συνεργασία με όλα αυτά τα συμπεράσματα και σήμερα εμείς αυτό που πρέπει να πούμε, ναι, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, πολλά ακόμα δεν τα έχουμε πετύχει, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε και αυτό είναι για μας πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Όπως είπατε, υπήρχαν τρία, τρεις κατηγορίες θεμάτων στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οποία αναφερθήκαμε με τους ε, αρμόδιους επιτρόπους ήταν και μία από τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, τους άξονες της Επιτροπής. Η Επιτροπή προχωράει σημαντικά στον τομέα της άμυνας. Οι προτάσεις της Επιτροπής σίγουρα στηρίχτηκαν ευρέως και εδώ έχουμε και τον Φιλίπ Μπρινέ, ο οποίος πλέον είναι θαμώνας της Επιτροπής μας. Θα μας μιλήσει σαν ειδικό θεμάτων ασφάλειας και άμυνας στον αεροδιαστημικό τομέα. Ποια είναι η ανάλυση σας των συμπερασμάτων αυτού του Συμβουλίου και πώς βλέπετε τις αποστολές της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Ντοζό. Να ευχαριστήσω την η Επιτροπή. Εισαγωγικά να σας πω μόνο ότι μιλήσατε για ένα ποτήρι μισογεμάτο ή μισό γεμάτο. Εμείς όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, το, την τρίτη κατηγορία, θα λέγαμε ότι το ποτήρι είναι μάλλον αρκετά γεμάτο. Για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε ένα πολιτικό και λειτουργικό τρίποδο. Μια δυνατή πολιτική ασφάλειας και άμυνας βασίζεται σε στρατιωτικές δυνατότητες που πρέπει να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην ενίσχυση και διατήρηση μιας βιομηχανικής τεχνολογικής βάσης σημαντικής και έρευνας. Δεύτερο σημείο το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι το Συμβούλιο έχει εκφράσει με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο την ενίσχυση και αυτό ξεκίνησε ήδη από τον Ιούλιο με την επικοινωνία της Επιτροπής και συμπληρώθηκε από προτάσεις που έκανε η Επιτροπή και που έχουν τεθεί σαν προτεραιότητες. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που θα αναφέρω εδώ, το οποίο μας υπενθύμησε ο Πέντρο και ο Μάτσακ, είναι το 2015 και η φιλόδοξοι στόχοι της συνάντησης κορυφής, φιλόδοξοι στόχοι που το 2008 εκφράστηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Τώρα, όσον αφορά πολύ συγκεκριμένα τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Πρώτον, η εσωτερική αγορά και οι δύο οδηγίες που υπάρχουν σήμερα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την υλοποίηση αυτών των ε, οδηγιών στην πλήρη τους διάσταση. Το πολιτικό μήνυμα των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ, ο Επίτροπος Ταγιάννη με τις οδηγίες εσωτερική αγορά και μεταφορά όπλων, εξοπλισμών η υλοποίηση λοιπόν αυτών των δύο οδηγιών σίγουρα προϋποθέτει πολύ ισχυρή πολιτική βούληση, κάτι που σήμερα δεν το έχουμε δει ακόμα πλήρως. Δεύτερο, είδατε ότι τα λέω όλα με πολύ πολύ προσεκτικό και διπλωματικό τρόπο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έρθηκε στην ασφάλεια του εφοδιασμού Κάτι που αποτελεί σημαντικό σημείο για μας και για την αμυντική συνεργασία και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Να προσθέσω εδώ, και εδώ αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάλερ, αλλά και στην έκθεσή του, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τρία θεσμικά όργανα που συνεισφέρουν για τους ίδιους στόχους. Δηλαδή, η διάσταση, η αμυντική διάσταση της εσωτερικής αγοράς δεν μπορεί πλέον να παραμελείται. Δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο από πολιτικής απόψεις είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη γενικότερη αρχιτεκτονική της βιομηχανίας εξοπλισμών. Το Συμβούλιο έχει υπογραμμίσει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βασιστούμε στις ανάγκες όπως έχουν παρουσιαστεί και εκφραστεί και να μην είμαστε προστατευτικοί καθότι σήμερα μία προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω μπορούν να εφαρμοστούν εδώ στους τομείς των εξοπλισμών, με την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι τα κοινοτικά εργαλεία δεν εφαρμόζονται μέχρι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την συνεισφορά τους. Αυτό σήμερα στον τομέα των εξοπλισμών μας οδήγησε σε μία εικόνα πολύ αποκλειστική σχέση κάποιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, κάποιων ε, μεγάλων ε, τομέων, κλάδων και επιχειρήσεων που σε περίπτωση παραδείγματος χάρη ε, κρίσης μειώνει δραστικά και αποφέρει πλήγματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραδείγματος χάρη στον τομέα του πολεμικού ναυτικού είναι οι κυρίοι πρωταγωνιστές. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πρώτες εταιρείες που πλήττονται είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, είναι η τυποποίηση και η πιστοποίηση. Οι δύο αυτοί τομείς έχουν αναγνωριστεί, εντοπιστεί από τους στρατιωτικούς, από την εξοπλιστική βιομηχανία και ο διαλειτουργικός χαρακτήρας, ο διεπιχειρησιακός χαρακτήρας πολλών επιχειρήσεων θα πρέπει μέσω μίας καλής διαδικασίας τυποποίησης και μίας διαφάνειας στην πιστοποίηση να μειώσει το κόστος τα εξοπλιστικά προγράμματα στοιχίζουν λιγότερο και η αγορά είναι πολύ πιο ευέλικτη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ σύντομα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, συζητήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τις υπάρχουσες διαδικασίες πιστοποίησης, τις διαδικασίες τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο και εδώ σκεφτούμε τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ βέβαια. Η πρώτη, αν θέλετε, διαδικασία, ο πρώτος στόχος είναι ο διαλειτουργικός χαρακτήρας. Και εδώ μπορούμε βεβαίως αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ να τα μεταφέρουμε χωρίς να τα υπονομεύσουμε και να κινητοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαργασίες, διαδικασίες, οργανισμούς ε, μη στρατιωτικούς θα τους χαρακτήριζα οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν για την ε, πιστοποίηση στον στρατιωτικό τομέα. Τέλος και ολοκληρώνω. Ο κύριος Σέλερ έφυγε, αλλά θα ήθελα να του πω ότι είναι σωστό να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχτηκε τα επόμενα χρόνια να ξεκινήσει μια προετοιμασία εντοπίζοντας την έρευνα στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για μια δράση προετοιμασίας, η οποία αν προχωρήσει σωστά, αν καθορίσουμε προσεκτικά τους στόχους, αυτή η προετοιμασία, η προετοιμασία σε τομείς όπου μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική κοινοτική δράση, αυτή η προετοιμασία είναι πάρα πολύ καλός τρόπος να φέρουμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια με μεγάλη επιφυλακτικότητα σε κάποιους άλλους τομείς όπως η ε, πολιτική προστασία, στον τομέα της πολιτικής προστασίας με εξαιρετικά αποτελέσματα και θυμάμαι τι επιφυλακτικότητα είχε προκαλέσει στην αρχή αυτή η πρόταση. Το ίδιο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε σήμερα για την ε, προετοιμασία της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας η οποία μπορεί να κινητοποιήσει το επόμενο κύκλο του δημοσιονομικού πλαισίου και να δούμε βεβαίως ποιο μπορεί να είναι και το περιεχόμενο. Κύριε Ντοζό, βεβαίως και θα προετοιμάσουμε εδώ ένα οδικό χάρτη, δεν τον έχουμε ακόμα ολοκληρώσει. Ελπίζω να είναι έτοιμο πριν το καλοκαίρι και υπό μορφή έκθεσης να υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε αυτό το έγγραφο θα προετοιμάσουμε τις δράσεις μας και τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν θα είναι μόνο τα κράτη, δεν θα είναι μόνο η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Δεύτερον, προτείναμε ο Επίτροπος Μπαρνέ και ο Επίτροπος Ταγιάννη, ο Πρόεδρος Ταγιάννη, θα συνεχίσουν με την Task Force Άμυνα και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης την προετοιμασία όχι μόνο του Συμβουλίου αλλά τον καθορισμό οι τρεις αυτοί φορείς θα κατανείμουν την εργασία μεταξύ τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει εδώ να παίξουν ένα ρόλο ο οποίος δεν θα αμφισβητείται. Οι δράσεις οι οποίες θα είναι προαιρετικές για τα κράτη-μέλη προϋποθέτουν την συμμετοχή των κρατών μελών αλλά και την ε, καθόλη τη διάρκεια της ε, επιχείρησης, συμμετοχή τους και διαβούλευση των κρατών μελών. Μηχανισμοί διαβούλευσης που προϋπάρχουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, διότι αυτό θα μας επιτρέψει και θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να στέλνουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον μη στρατιωτικό τομέα και οι οποίοι θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να αξιολογήσουν αυτά που συμβαίνουν ε, στις νέες επιχειρήσεις ολοκληρώνω με μια πρόσκληση. 4 Μαρτίου οι δύο επίτροποι Μπαριέ και Ταγιάννη θα οργανώσουν μια συνδιάσκεψη για την προετοιμασία του οδικού χάρτη και εξ ονόματος του Αντιπροέδρου Ταγιάννη και του Επιτρόπου Μπαρνιέ σας προσκαλώ όλα τα μέλη της Επιτροπής σε αυτήν την συνάντηση. Ευχαριστούμε για αυτήν την διεξοδική και λεπτομερέστατη παρουσίαση θα έλεγα για να οργανώσουμε σωστά τη συζήτησή μας να ακούσουμε ευθύ αμέσως τον ε, κ. Τουλέα, ο οποίος είναι μόνιμος εκπρόσωπος στην ε, Επιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας. Ε, φαντάζομαι ότι θα μας πούν οι ειδικοί νομικά, ότι δεν υπάρχει προεδρία για τα θέματα αυτά, εναλλασσόμενη προεδρία, όμως για μας σε θέματα πολιτικής, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξέρετε καλύτερα τις προτεραιότητες που πρέπει να προωθηθούν και υπό το φως των όσων υπόθηκαν, θέλουμε να δούμε τι συνέχεια θα λάβουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Θα είναι σίγουρα πολύ πολύμορφη η υλοποίηση των στόχων αυτών. Και βεβαίως η Ελλάδα θα υποδεχτεί το επιτελείο της μελλοντική επιχείρησης στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Οπότε η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα για, το, για την Ένωση τους ερχόμενους έξι μήνες θα έχει να διαρματίσει ενεργότατο ρόλο. Με χαρά λοιπόν να σας ακούσουμε. Uh, thank you very much. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και εγώ είμαι έτσι αυστηρός ε, ε, περί τα νομικά ειδικό. Ξέρουμε ποιος είναι ο θεσμικός μας ρόλος ε, και θα τον φέρουμε σε πέρας με τη δέωση επιμέλεια. Αξιότιμοι βουλευτές κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο η πρόσκληση που μου απευθύνεται να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση και να παρουσιάσω την προοπτική των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το μέλλον της ΚΕΠΑ. Η... Από τη Ελλάδα, βέβαια, που πάντα ήταν υπέρμαχο μια ισχυρότερη ε, συμμετοχή και ενό ισχυρότερου ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη ασφάλεια και άμυνα. Πρέπει να αναλάβουμε τη διεθνή μα ευθύνη στον τομέα τη ασφάλεια. Δεν είναι πλέον επιλογή, είναι αναγκαιότητα κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα επηρεάζεται και λόγω των εξελίξεων των εσωτερικών, ε, ιδίως στη γειτονική περιοχή, Ανατολική Μεσόγειο, μεταναστευτικές ροές, αστάθεια. Αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Επίσης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πλήρες δυναμικό, της δυνατότητες που μας προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας ιδίως σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΑ. Παραδοσιακά είμαστε υπέρμαχος ενός ενισχυμένου λοιπόν ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θεωρούμε ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να αποφαίνεται φόλων των πολιτικών μεταξύ αυτών και της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑ. Επίσης, αξιολογούμε την ε, συνεισφορά των κρατών μελών, μάλλον του Κοινοβουλίου υπό μορφή εκθέσεων. Ενδεικτικά να αναφέρω την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου, της κυρίας Κοπά και της κυρίας Κόμες που είναι και παρούσα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πολύ αναμενόμενο γεγονός, υψηλές προσδοκίες. Πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς θα θέλαμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι στον πιο φιλόδοξο για να εκπέμψουν ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα. Αξιολογούμε το αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι ακρογωνιαίοι λύθοι που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η άμυνα πλέον θεσμικά θα έχει συνέχεια, δεν θα είναι κάτι που γίνεται άπαξ. Θα υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Θα είναι συνεχώς λοιπόν ε, στο θεματολόγιό μας και πρώτη φορά στην Αθήνα 20 και 21 Φεβρουαρίου που έχουμε την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας και βέβαια αργότερα τον Απρίλιο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην δυνατότητά μας να δρούμε από μόνοι μας ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Και θέλουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος πάροχος ε, ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να τονίσουμε επίσης ε, το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των ε, συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας, και το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών που συνεισφέρουν στη δημιουργία μια κοινή κουλτούρα νοοτροπία όταν τη ασφάλιση τη άμυνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ειδικό ρόλο που, ανέφερε ο πρόεδρο, εφόσον έχουμε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εξάμεινο, διαφορετικός ρόλος αυτός βέβαια, σε σχέση με την εποχή πριν τη Λισαβόνα. Εμεί θέλουμε να εφαρμόσουμε τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενεργά, στηρίζοντα ε, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την ΕΙΕΔ. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την εκπόνηση και την υλοποίηση μια στρατηγική θαλάσσια ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε να εγκριθεί η σχετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014. Επιπροσθέτως, άλλοι τομεί ε, ενδιαφέροντο. Είναι η κυβερνοασφάλεια, βιωσιμότητα στην άμυνα, ανάπτυξη ικανοτήτων και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Βάση. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις ε, ικανότητές μας, να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων με τη διασύνδεση δυναμικών βιομηχανικών τομέων και με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ε, προανέφεραν και οι άλλοι ομιλητέ, η εταίροι είναι ένα στοιχείο κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, η Ηνωμένα Έθνη και άλλες οργανώσεις. Και βέβαια μεταξύ αυτών πολύ σημαντικό είναι να έχουμε και στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ έτσι ώστε να, αποφα... Ε, να, αποτρέ... να αποφύγουμε τις και να χρησιμοποιήσουμε ε, με τον πλέον σόφρονο τρόπο τις ικανότητές μας. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία επίσης με βάση μια πραγματική οργανωτική προσέγγιση. Αλλά να υπάρχει και αυτονομία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, σφαιρική προσέγγιση, αυτή το comprehensive approach. Είδα ότι πολύ ενδιαφέρεστε για το θέμα αυτό, την διαχείριση κρίσεων, τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε προκλήσεις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την κοινή ανακοίνωση ΕΕ και Κομισιόν σε σχέση με τη σφαιρική αυτή προσέγγιση, τη συνολική προσέγγιση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Merci, monsieur euh, Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκόμες. Ε, Έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο παρεμβαίνοντες για τις ομιλίες τους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το Συμβούλιο και θα ήθελα να απευθυνθώ στον, στην Ελληνική Προεδρία τώρα. Εάν δεν το έκανε το Συμβούλιο θα πιέσει η Ελληνική Προεδρία να γίνει απολογισμός των συνεπειών, των επιπτώσεων στις ε, χώρες όπου υπάρχει πρόγραμμα της Τρόικας και τις δικές τους ε, συστάσεις, τις δικής τους βιομηχανικής βάσης για την άμυνα διότι γνωρίζοντα την κατάσταση τη δική μου χώρα, ε, η κατάσταση, ο αντίκτυπο είναι καταστροφικό. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό τουλάχιστον και να ε, λάβει διορθωτικά μέτρα. Εάν είμαστε σε διαδικασία διάσωση, εμεί στην Πορτογαλία, ίσω και εσεί στην Ελλάδα και άλλοι, αυτό είναι επειδή υπήρχε πολλή διαφθορά. Και σίγουρα υπήρχαν πολλέ δαπάνε, υπέρμετρε δαπάνε, στι οποίε. Ε, περάσαμε και εμείς ε, στη χώρα μας λόγω των μακρονομικών ανοσυροποιών, λόγω του ευρώ, ε, του φτηνού ευρώ, όμως οι κρατικές δαπάνες ήταν κυρίως δαπάνες στην άμυνα και σε ένα πλαίσιο διαφθοράς. Με πραγματικά με μια σειρά από επεισόδια διαφθοράς. Να θυμίσω την υπόθεση των υποβρυχίων. Ξέρω ότι και στην Ελλάδα ε, ψάχνετε ακόμα την αλήθεια και τους υπεύθυνους για αυτήν την περίπτωση, αλλά πουθενά στη χώρα μου δεν υπήρξε μια σύμβαση άμυνας και ασφάλειας τα τελευταία χρόνια που να μην υπάρχει διαφθορά αλλά και που να μην εμπλέκονται χώρες από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι διαφθορά λοιπόν στην Πορτογαλία αλλά στους απέναντι. Αυτό πραγματικά αποδυναμώνει το στρατιωτικό μας δυναμικό και την όλη μας προσπάθεια και την εικόνα μας στην κοινή γνώμη αλλά δείτε τι γίνεται εκεί που υπάρχουν σαφείς επιπτώσεις. Η σύμβαση αυτή για τα υποβρύχια ε, έγινε το 2002. Ήταν ο Πρωθυπουργός ο κ. Μπαρόζο, ο τωρινός ε, ε, ε, υπουργός αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία ήταν υφυπουργός άμυνας. Υποτίθεται ότι τα υποβρύχια κόστησαν ε, περίπου 100 εκατομμύρια και τελικά ε, η τιμή που πληρώθηκε ήταν ένα δις περίπου. Το 52% υποτίθεται ότι θα πηγαίναν στα ναυπηγεία του, της ε, πόλης Βιάννα του Καστέλου, που είναι τα μόνα ναυπηγεία που φτιάχνουν σκάφη για το ναυτικό μας. Εκεί κατασκευάζονται τα σκάφη του πολεμικού μας ναυτικού. Προφανώς αυτά τα κέρδη έπρεπε να γίνουν ε, εντολές, μεταφορά τεχνολογίας, μεταφορά εξοπλισμού. Ήταν ο εξοπλισμός λοιπόν που πωλήθηκε, υπερτιμημένος, εντολές δεν πέρασαν όπως είχε υποσχεθεί και καμία μεταφορά τεχνολογίας δεν έγινε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, η τερνική κυβέρνηση λέει ότι δεν έχουν αξία πλέον αυτά τα ναυπηγεία από μόνα τους και επινοικιάζουν, επιμισθώνουν αυτά τα ναυπηγεία μαζί με το λιμάνι, ένα από τα σημαντικότερα της Πορτογαλίας. Οπότε όχι μόνο καταστρέφεται η ναυπηγική μα βιομηχανία που παρήγαγε για το δικό μας πολεμικό ναυτικό σκάφι, <clears throat> αλλά θα έχουμε και άλλα μπλεξίματα στο εξωτερικό, με άλλα βρώμικα χρήματα, με άλλα ε, κέρδη ε, που δεν θα αποδοθούν σε αυτούς που πρέπει, αλλά όχι μόνο αυτό. παραχωρούμε ένα λιμάνι που είναι πολύ σημαντικό για την ειδική μας την άμυνα σε μια εταιρεία που δεν δίνει καμία εγγύηση ότι θα ε, πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους. Για να μην πω καν για την κατασκευή σκαφών. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα πόσο καταστροφικά είναι όλα αυτά. Τι είναι λοιπόν όλη αυτή η κουβέντα για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης προς όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στις χώρες όπου επιβάλλεται πρόγραμμα λιτότητα με τέτοιες φιλελεύθερες πολιτικές. Όχι, εδώ αποδεκατίζουμε τις δυνατότητές μας και νομίζω ότι πραγματικά τραυματίζουμε χώρες όπως η δική μου ενώ υπήρχαν βασικά στοιχεία για να παράγουμε αυτά που τώρα απαγγέλουμε και αναγγέλουμε στόχους. Επίσης, θα ήθελα να σκεφτούμε το εξής. Κατά πόσον χάνουμε τον έλεγχο των δυνατοτήτων μας, ιδίως των τεχνολογικών, όταν όλα, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας είναι προς πώληση και μάλιστα μισοτιμής για τους Κινέζους. Είναι λία στα χέρια των Κινέζων και χάνουμε τις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και σε αυτό το τομέα. Για να σκεφτούμε λίγο τι χάνουμε, τι δυνατότητες χάνουμε και να μην αναφέρω και πάλι τον έλεγχο των στατογικών σημείων της ε, επιτρατείας μας της Αφρικατής της Ευρώπης. Μίλησα για το ευαίσθητο λιμάνι της Βιάννα του Καστέλου. Τι γίνεται με το λιμάνι του Πειραιά και την κινέζικη εταιρεία που μισθώνει. Πιέζει την Ελλάδα να πωλήσει πλήρως στην περίπτωση, στη χώρα μου λόγω χάρη, έχουμε δύο, μία βασική μάλλον εταιρεία παραγωγό ενέργειας για το ηλεκτρικό και για την ε, παροχή ηλεκτρικού. Παλιότερα είχαμε κάνει αποσύνδεση της παραγωγής και της ε, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από ε, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά με τις ευλογίες της Τρόικας σε ποιους πολίθηκαν αυτές οι εταιρείε στους ε, Κινέζους, σε εταιρείες που ελέγχονται από το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τι μου λέτε, η ενέργεια δεν είναι στρατηγικό ε, περιουσιακό στοιχείο, όχι μόνο για την Πορτογαλία, αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κανείς δεν κάνει τίποτα. Πού είναι η λογική όλων αυτών. Τι μιλάμε για βιομηχανική βάση για την άμυνα. Εάν πραγματικά όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει σε αυτήν την δημιουργία. Κύριε Γκάλερ. Λίγο πιο σύντομα αν γίνεται. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Επειδή είναι εδώ ακόμα ο κύριος ε, Σεράνο, ακούσαμε κάποια τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και το ερώτημα είναι ποιος θα συνεχίσει. Θα επανέλθει του χρόνου, τον Ιούνιο, το Συμβούλιο για την παρακολούθηση και την υλοποίηση αυτών των ε, στόχων ή κάποιοι συνδυασμοί θεσμικών οργάνων, για να το πω έτσι, θα παρακολουθήσουν και θα υλοποιήσουν. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν όσον αφορά την προετοιμασία και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να υπάρξει αυτή η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα υπάρξει παραδείγματος χάρη η χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών ε, με μεικτή χρήση, στρατιωτική και μη στρατιωτική. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες που θα προχωρήσουν. Επίσης το θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού. Αυτό και τι δεν προχώρησε. Ποιες είναι οι αιτιολογήσεις. Μπορεί να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε το θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι εγγυήσει εδώ πρέπει να δοθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μπρινέ θα απαντήσει. Θα ξεκινήσω με τον έλεγχο των επενδύσεων και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εδώ υπάρχουν πάρα πάρα πολλές, πολλά ερωτηματικά και πολλές αιτίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να κατανοήσουμε γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Εάν είναι το ίδιο και έχει την ίδια έκταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και με τον κλάδο, δηλαδή τη βιομηχανία των εξοπλισμών. Όσον αφορά λοιπόν την ασφάλεια του φουδιασμού, πιστεύω ότι πρέπει, όπως αποφασίσαμε, να ξεκινήσουμε με μια νέα πρωτοβουλία με στόχο να καθοριστεί το εύρος του προβλήματος. Εδώ υπάρχουν ε, διάφορες ε, πιθανές διαμάχες μεταξύ των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και αυτών που θα ήθελε να εκτελέσει η Επιτροπή. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, κύριο Ποπόφσκι σίγουρα ξέρει καλύτερα το θέμα από μένα, αλλά πρόκειται για ένα παράδειγμα καλό που θέλει να εξετάσει η Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες και για λόγους στρατιωτικούς και για αποστολές στρατιωτικές αλλά και για μη στρατιωτικές αποστολές. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον εξοπλισμό με διπλό τρόπο. Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος και όχι ο Αντιπρόεδρος Τελιάννη, καθότι η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, τις κρατικές προμήθειες. Εδώ ζητούνται απαράδεκτα αντισταθμιστικά, τα οποία πραγματικά είναι αντίθετα με το πνεύμα της ε, και όπως είπατε πολύ σωστά, όλες οι μελέτες μας δείχνουν σήμερα ότι δεν υπάρχει οικονομική λογική, ότι υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού, ότι αυξάνεται το κόστος των εξοπλισμών και μπορεί πολύ βραχυπρόθεσμα να θεωρηθούν ενδεχομένως ε, πλεονεκτήματα. Μακροπρόθεσμα όμως πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό εμπόδιο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και για τα δύο αυτά παραδείγματα και τις κρατικές προμήθειες αλλά και την περίπτωση της μεταφοράς εξοπλισμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελών θα πρέπει να εξεταστεί. Και από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ αυτή η οδηγία, πολλά κράτη-μέλη έχουν καταργήσει ή έχουν αναθεωρήσει την νομοθεσία τους για το θέμα αυτό. Όπως σας έλεγα όμως στην αρχή όταν πήρα το λόγο, χρειάζεται εδώ και μια πολιτική βούληση. Η Επιτροπή πρέπει να την δείξει έτσι ώστε αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη να απαγορευθούν. Ε, thank you very much. well... Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος και πραγματικά είναι αφοσιωμένο στον, ε, στις ενόπλες δυνάμεις του και είναι πρόθυμος να πληρώνει φόρους για να έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ισχυρό στρατό. Η χώρα μας έχει μια διαρκή απειλή για πόλεμο από γείτονα χώρα, ιδίως ως προς το κάποια δικαιώματά μας ε, για τα διεθνή χωρικά μας ύδατα. Ε, ναι, υπήρξε διαφθορά, αλλά αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι, οι ιατουργοί βρίσκονται στη φυλακή, υπάρχει ενεξελίξη έρευνα και ανάκριση και είναι μια διαδικασία που προχωρεί. Όσο για τις συναλλαγές με την Κίνα, καμία χώρα πια στον κόσμο δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτό. Όλοι έχουν ε, εμπορικές σχέσεις με την Κίνα για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και για το τερματικό του Πειραιά, ναι, έχουμε σχέσεις με την Τουρκία. Με, συγγνώμη, με την Κίνα. Κύριε Σεράνο, ναι, μια πολύ άμεση απάντηση για το Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει σκοπό να συνεχίσει να προωθεί αυτή τη διαδικασία και αν χρειαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προκαλεί συζήτηση για όλα αυτά προκειμένου να προχωρήσουν τα διάφορα θέματα όπως η συνθήκη για πρώτη συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης για θέματα όπως εξοπλισμός, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ζητήθηκε από την είπατε εκπρόσωπο να εκπονήσει πολύ σύντομα προτάσεις. Υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα και στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε τον Πρόεδρο θα τα φέρνουμε αυτά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάντως συνεχίζουμε να βγαζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους της ΕΕΔ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και φυσικά θα διατηρήσουμε αμύωτη τη συμμετοχή μας. Έπειτα το 2015 και πάλι έχουμε ένα μεγάλο ραντεβού. Ένα ραντεβού που όπως ξέρετε θα συνοδευτεί από έκθεση του Συμβουλίου. Έκθεση από την οποία θα επωφεληθεί, θα, στην οποία μάλλον θα συμπεριληφθούν οι ε, πολύτιμες συνεισφορές της ΕΕ της και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να διευκολύνουμε λοιπόν την υλοποίηση και αν προκύψουν δυσκολίες θα προσπαθήσουμε να τις διαλύσουμε. Merci. Pas d'autres euh, interventions. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον πρέσβη, τον Γενικό Διευθυντή. Κύριε Σεράνο, σας ευχαριστώ. Έχετε σαλιγκάρια στην γραβάτα σας. Εγώ είμαι από την Βουργουνδία. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό αναφέρεστε με τα σαλιγκάρια και όχι στην ταχύτητα εξέλιξη της πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Ποχόφσκι. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση. Η ΜΕΝ και η ΔΕ έχουμε ενδεχομένως διαφορετικές θέσεις για το θέμα αυτό. Παρόλα αυτά, περιμένουμε να εξελιχθεί η κατάσταση και σαφώς και θα παίξουμε το ρόλο που μας περιγράψατε, να πιέζουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας για να κατευθυνθούμε όλοι στην σωστή κατεύθυνση. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπε ο Μικαέλ όσον αφορά τα μία πανδρομένα αεροσκάφη και τη χρησιμοποίησή τους σε μη στρατιωτικές αποστολές. Και όλοι μαζί με την υπηρεσία άμυνας και με τον επικεφαλής των στρατηγό Ντερουζιέ θα ακούσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί στις 9 και θα μιλήσουμε για την δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής.